Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous propose de faire silence et d'ouvrir nos travaux. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σε εργασίε μα θα ήθελα να καλωσορίσω όλου του συμμετέχοντε τη Ειδική Επιτροπή για την Φορολογία με την παρουσία ε, μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων, θα ήθελα επίση να καλωσορίσω τον εκπρόσωπο της Ολλανδικής ε, Προεδρίας. Πρόεδρο της ε, Επιτροπής Οικονομικών Αποθέσεων του Ολλανδικού ε, Κοινοβουλίου. Καθώς επίσης και όλους τους εκπροσώπους των 20, από 20 χώρες των κοινοβουλίων που παρίστανται από 30 κοινοβουλευτικά σώματα θα ε, είχαμε ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση εάν υπήρξαν κάποια μικρά προβλήματα, όπως για παράδειγμα το γεγονό ότι σε κάποιες ε, χώρες ε, ε, ε, ε υπήρχαν ξανακλογέ πρόσφατα, ενώ άλλοι εκπρόσωποι δεν μπόρεσαν να έρθουν εξαιτία των τραγικών επιθέσεων που όλοι γνωρίζουμε στο αεροδρόμιο του Ζάβιντερ. Το πρώτο σημείο τη τη διάταξη είναι η υιοθέτησή τη. Το δεύτερο σημείο είναι οι ανακοινώσει του Προέδρου. Η συνεδρίασή μα είναι δημόσια, όπω και όλε τι συνεδριάσεις τη Ειδική Επιτροπή μα. Ε, μεταδίδεται και μέσω web streaming στο ίντερνετ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να ακούσετε και να ομιλήσετε και τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως βλέπετε εγώ μιλώ γαλλικά, μπορείτε και εσείς να μιλήσετε τη γλώσσα σας. Θα ήθελα απλώς να επενθυμίσω ότι έχει παραταθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου η θητεία της Επιτροπής μας. Τα πρώτα συμπεράσματα δημοσιοποιήθηκαν το Δεκέμβριο της προηγούμενου, προηγούμενου έτους και τα τελικά συμπεράσματα μας θα τα παρουσιάσουμε τέλος Ιουλίου. 28 Απριλίου επίσης να σας επιθυμίσω ότι οργανώνουμε ε, μια συζήτηση επί εκθέσεων που εκπώνησε το Τμήμα Πολιτικής, η Διεύθυνση Α, και επίσης να σας ενημερώσω ότι πρόκειται να διοργανωθεί ακόμα μια συνάντηση με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και των 28 κρατών μελών αλλά επίσης και οι εκπρόσωποι κοινοβουλίων των 80 κρατών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του ΟΣΑ για την υιοθέτηση των κανόνων BEPS. Πολύ σύντομα σε λίγες εβδομάδες θα διοργανωθεί αυτή η συνάντηση στο Παρίσι και θα έχουμε τη δυνατότητα, αφού θα έχουμε ήδη ανταλλάξει μεταξύ μας στους ευρωπαϊκές χώρες τις ε, απόψεις μας, να τις εκφράσουμε αυτές και προς τους εκπροσώπους των υπολείπων ε, χώρων που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ λοιπόν στο επόμενο σημείο ε, θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά των προηγούμενων δύο συνεδριάσεων θα θεωρήσω ότι ενεκρίθησαν εάν δεν εκφραστεί κάποια επιφύλαξη, κάποια διόρθωση μέχρι το τέλος της συνεδρίας. Λίγα λόγια για να υπενθυμίσω ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής συνάντησης και το πλαίσιο εντό του οποίου τη διοργανώνουμε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πίτερ Βέζερμπερκ, τον πρόεδρο της μόνιμης Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του ε, Κοινοβουλίου της Ολλανδίας. Δυστυχώς δεν θα μπορέσει να μείνει μαζί μας στο τέλος της ε, συνάντησης, αλλά θεωρώ την παρουσία του πολύ σημαντική. Μιας και εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο ε, της χώρας που έχει αναλάβει την ε, Προεδρία του Συμβουλίου και θα συμπροεδρεύσουμε σε αυτήν τη συνάντηση σήμερα ένας εκπρόσωπος από την Ολλανδία λοιπόν και ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης να ενημερώσω ότι από τα 20 κοινοβουλία που εκπροσωπούνται σύντομα, ε, ε σήμερα εδώ, τα 10 εκπροσωπούνται στο επίπεδο του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Προϋπολογισμού ή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους 5 λεπτά ο καθένας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Γαλλικό Κοινοβούλιο, καθώς επίσης και α, τους εκπροσώπους των της των Κοινοτήτων του ε, Ηνωμένου Βασιλείου που μας απέστειλαν γραπτές παρατηρήσεις και με την ευκαιρία να πω και σε όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ παρόντος ότι μπορούν να αποστείλουν και εκείνοι γραπτά σχόλια. Ποια είναι η γενική ιδέα. Τι προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα. Θέλουμε να αντιληφθούμε ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις των Εθνικών Κοινοβουλίων ως προς τις διάφορες προτάσεις που έχουν κατατεθεί για τον τρόπο με τον οποίο θα καταπολεμήσουμε την φοροαποφύγη των επιχειρήσεων, αυτές οι προτάσεις οι οποίες έχουν ε, κατατεθεί τους τελευταίους 18 μήνες. Και έχουμε διάφορα σκάνδαλα που συνέβησαν τους τελευταίους αυτούς μήνες, αρχικά Leaks και πρόσφατα, πιο πρόσφατα ε, τα έγγραφα του Παναμά, Panama Papers, που μας δείχνουν πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, το οποίο εμείς θα πρέπει να καταπολεμήσουμε έτσι ώστε να υπάρξει μια σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, με, χωρίς τρευλώσεις του ανταγωνισμού, κάτι το οποίο είναι σημαντικό επίσης και για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας την ε, παγκόσμια οικονομία. Ο ΩΣΑ και η G20 έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες την τελευταία χρονιά. Η πρώτη σχετική απόφαση είχε ληφθεί ε, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από Λουξεμβουργιανής Προεδρίας. Ήταν η απόφαση για την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τις αποφάσεις ε, φορολογικές, tax rulings. Και Μετά έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αυτή τη στιγμή εξετάζεται υπό Ολλανδικής Προεδρίας στο Συμβούλιο. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά προτάσεων που σας έχουμε αποστείλει. είτε πρωτοβουλίε οι οποίε αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω για παράδειγμα ένα αρμόνιση του φορολογικού καθεστώτο των μεγάλων επιχειρήσεων, ή επίση ε, πρωτοβουλίε σε παγκόσμιο επίπεδο, τι οποίε παρακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τη του ΟΣΑ. Το δεύτερο εξάμεινο του έτους αναμένουμε και τη σχετική πρόταση του πακέτο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η φορολογία είναι εθνική αρμοδιότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα, είναι δική σας αρμοδιότητα λοιπόν των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αλλά με επί ευκαιρία συναντήσεων όπως η σημερινή, μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις, ιδέες, την αξιολόγηση του καθένα μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη και η ευρωπαϊκή και η διεθνής διάσταση στις εθνικές αποφάσεις που τελικά θα λαμβάνονται. Βεβαίως κάθε χώρα αποφασίζει η ίδια. Και στο βαθμό που υπάρχουν η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάλι ε, οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία επομένως θα μπορούσαν να λοκαριστούν σε περίπτωση που ένα κοινοβούλιο με κυβέρνηση ή ακόμα και ένα δημοψήφισμα ε, της ε, ε, σταματούσε. Αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε στη συμφωνία, τη μέγιστη δυνατή συμφωνία που μπορούμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε επίσης να παρουσιάζουμε μια κοινή θέση έναντι των συνομιλητών μας στον ΟΣΑ. Μέσα Μαΐου έχουν γίνει επαφές με τον Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών έτσι ώστε να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων και να έχουμε την ίδια ε, θέση ή δυνατόν να συμφωνήσουμε ε, σε κοινέ θέσεις ε, για την κατεύθυνση που θα πάρει η πρωτοβουλία του ΟΣΑ. Θα δώσω αμέσως τον ε, λόγο στον κύριο Πίτερ Τουίσπερκ για να μας κάνει μια μικρή παρουσίαση. Μετά στον κύριο Στίβεν Κουέστ, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του εδώ που θα μας παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Και μετά, όπως σας είπα, θα δώσουμε το λόγο για πέντε λεπτά στον καθέναν από τους τέσσερις προέδρους ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών που μας τίμησαν με την παρουσία τους, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, από τη γερουσία της Ιταλίας, ε, από τη γερουσία της Πολωνίας. Και μετά θα δώσουμε το λόγο ε, εναλλάξει σε έναν ε, εκπρόσωπο Εθνικού Κοινοβουλίου και σε έναν Ευρωβουλευτή. Έχετε τη σχετικά έντυπα για να ζητάτε το λόγο. Ο κύριος Ντουίσπερκ. Σας ευχαριστώ κύριε Λαμασούρ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Αλένα Μασούρ για την ε, διοργάνωση αυτής της συνάντησης με τα Εθνικά Κοινοβούλια και για την πρόσκλησή του για να κάνω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Στη διάρκεια του γεύματος είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων για το κεντρικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Είναι ήδη προφανές ότι είναι πολύ επίκαιρη αυτή η συνεδρίαση γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους τελευταίους μήνες και εβδομάδες έχει δημοσιεύσει πολλές ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα. Αλλά έχουμε και τις πληροφορίες για τα έγγραφα του Παναμά, το Panama Papers, το σκάνδαλο. Και σήμερα συζητούμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν υπάρχει ούτε μία βουλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τα θέματα της φορολογίας και οι πρόσφατες εξελίξεις δεν βρίσκονται στο, στην πρώτη σελίδα της σας τους διάταξης. Και μάλιστα ε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω και εγώ τις παρατηρήσεις μου για τις ε, δράσεις και τις απόψεις της ε, Ολλανδικής Κυβέρνησης και τις ε, δράσεις της Ολλανδικής Βουλή των Αντιπροσώπων. Καταρχήν, προς προ την θέση της Ολλανδικής Κυβέρνησης. Στην επιστολή τη Δευτέρα Ιουνίου 2015, η Ολλανδική Κυβέρνηση υιοθέτησε μία σαφή θέση στο θέμα τη αντιμετώπιση της ε, φοροαποφυγή κυρίω πολυεθνικών ομήλων. Ε, θέλουμε να διατηρήσουμε ένα πρόσφορο ε, ταυτόχρονα επενδυτικό κλίμα για τις επιχειρήσεις. Η Ολλανδική κυβέρνηση θέλει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΣΑ προκειμένου να παταχθεί η φοροαποφυγή. Μάλιστα στην επιστολή η κυβέρνησή μας ε, ανέφερε σε ποιους τομείς θα ήθελε να πρωτοστατήσει. Συγκεκριμένα θα ήθελε να ενισχυθεί η διαφάνεια για παράδειγμα στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φοριών και των φορολογικών συμφωνιών τύπου tax rulings μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων. Επίσης θέλουμε να ε, ενισχύσουμε τις κατευθυντήρες γραμμές του ΩΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης. Και επίσης ό,τι αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, ε, θέλουμε να τροποποιήσουμε υπάρχουσες φορολογικές συμφωνίες προκειμένου να ενισχυθεί το, ενισχυθεί το δυναμικό των δικών τους φορολογικών διοικήσεων. Επίσης, θα πρέπει να πατάξουμε τις καταχρήσεις σε, πολ... σε διεθνές επίπεδο, πολυμερές επίπεδο, με σκληρό δίκαιο. Για παράδειγμα, έχουμε καταχρήση συνθήκων, προνομιακά, φορολογικά καθεστώτα, φορολογικές συμφωνίες. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε την σχετική μας πολιτική μέσω ενός δικτύου, αλλά και εκ των προτέρων να αντιμετωπίσουμε αυτές τις φορολογικές συμφωνίες τύπου tax rulings. Μετά την υιοθέτηση της έκθεσης BEPS του ΟΣΑ στις 5 Οκτωβρίου, η Ολλανδική κυβέρνηση διατράνωσε και πάλι την υποστήριξή της. Ε, θέλουμε κοινά προδιαγραφές εκθέσεων και αυτό με την ταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και επίσης είμαστε υπέρ των εκθέσεων αναχώρα. Και μάλιστα ως ε, ασκώντας την Προεδρία ε, θέλουμε να αναζητήσουμε συμβαστικές λύσεις και να βρούμε συμβαστικές προτάσεις για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ε, για να λαμβάνουμε αποφάσεις και να διατηρήσουμε συνθήκες ίσου ανταγωνισμού διατηρώντας ένα πρόσφορο επενδυτικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Ποιε είναι τώρα οι αντιδράσει της Ολλανδικής Βουλής των Αντιπροσώπων. Η κάτω βουλή της Ολλανδίας έχει θετήσει πολλές ε, θέσεις, κατά πλειοψηφία μάλιστα. Θα επικεντρωθώ σε έξι προτάσεις που εθετήθηκαν στην Ολλανδική Βουλή και που ίσως απτώνται ε, ε, και της απογευματινής αυτής της συζήτησης. Καταρχήν, η Κάτω Βουλή της Ολλανδίας παροτρύνει την κυβέρνηση να αναπτύξει ένα σχέδιο και να διατηρήσει την ελκυστικότητα του Ολλανδικού επενδυτικού κλίματος για τις διεθνείς επιχειρήσεις με υπεύθυνο όμως τρόπο. Δεύτερον, η Βουλή των Αντιπροσώπων των Κατοχωρών ζήτησε από την κυβέρνηση να διαχωρίσει το πακέτο, τη δέσμη μέτρων ΑΤΑΠ για την πάταξη φοροαποφυγή σε δύο σκέλη. Στο σκέλο ΩΣΑ και στο σκέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που ευθυγραμμίζεται με την πρόταση τη Γερμανία στο Συμβούλιο Εκοφήν τη 12η Φεβρουαρίου. Τρίτον, η Ολλανδική Βουλή ζήτησε μελέτη επιπτώσεων των διαφόρων ε, συνιστοσών της οδηγίας κατά της διάβρωσης βάσης και μετατόπισης κερδών ε, με βάση τις προτάσεις της Φιλανδίας, Λουξεμβούργου, Βελγίου και άλλων χωρών στο ίδιο κοφήν της 12ης Φεβρουαρίου. Τέταρτον, η Ολλανδική Βουλή ζήτησε από την κυβέρνηση να προσπαθήσει να καταλήξει συμφωνία για τη δέσμη μέτρων για την πάταξη της φοροαποφύγη στο ΑΤΑΠ, μάλιστα σε αυτό το εξάμεινο, κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας. Πέμπτον, ενίσχυσαμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης να ε, ε, υιοθετηθούν πανευρωπαϊκές ε, εκθέσεις αναχώρα και επίσης ενισχύουμε τις κυβερνητικέ ε, ε, προσπάθειες ε, να δημιουργηθεί μια μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συναφών δικαιοδοσιών. Αυτέ λοιπόν ήταν οι απόψει και αντιδράσει τη Ολλανδική Βουλή. Τέλο, λίγα λόγια για τα έγγραφα του Παναμά, πολύ πρόσφατα. Τα έγγραφα του Παναμά δεν αφορούν πολυεθνικού ομίλου, αλλά συγκεκριμένου ιδιώτε, φυσικά πρόσωπα, ε, που μετατόπισαν τα περιουσιακά του στοιχεία εκεί. Βέβαια, διαφάνεια δεν υπάρχει, έτσι φαίνεται, και αυτά τα περιουσιακά ε, στοιχεία δεν έχουν αναφερθεί στις αρμόδιες φόρειες, Κάτι που ίσως ε, οδηγεί σε φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή που είναι αξιόπινη πράξη και αυτό προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πρόσφορο επενδυτικό περιβάλλον για τις διεθνείς επιχειρήσεις. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να εκφράσω και πάλι την πεποίθησή μου ότι αυτό που προέχει σήμερα είναι να διδαχθούμε ο ένας από τον άλλον και να προωθήσουμε τη διεθνή συνεργασία μεταξύ μας. Αυτό είναι ζωτική σημασία, γιατί τα φορολογικά συστήματα δεν προσαρμόζονται στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο ε, των αγαθών και υπηρεσιών. Γι' αυτό μόνο με συνεργασία μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστούμε για τα πολύ συγκεκριμένα σχόλιά σας και τις απόψεις της Ολλανδικής Βουλής που μας μεταφέρατε πιστά. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Στίβεν Κουέστ, το Γενικό Διευθυντή της Αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Λαμασού. Με ιδιαίτερη ευτυχής για την πρόσκληση που με απευθύνατε να συζητήσουμε μαζί το ζήτημα της φορολογικής ε, δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα το ζήτημα της καταπολέμησης της φοροαποφυγής από επιχειρηματικούς ομίλους και ιδιαίτερα από επιχειρήσεις. Και σε αυτό θα εστιάσω. Βέβαια, δεν θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει τη συζήτηση χωρίς να αναφερθεί στο σκάνδαλο των εγγράφων του Παναμά, του Panama Papers. Και θα ήθελα γι' αυτό το λόγο να κάνω κάποιες σχετικές παρατηρήσεις πρώτα. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι τα έγγραφα του Παναμά μας δείχνουν πόσο απαραίτητη είναι η συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση τη φοροαποφυγή. Εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζουμε, να δημιουργούμε ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και όσον αφορά τους ατομικούς λογαριασμούς και όσον αφορά την πραγματική κυριότητα και την καταπολέμηση της, ε, της νομοποίησης ε, εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όμως αυτό θα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς προσπαθούμε να ε, πιέσουμε και τρίτες χώρες σε διεθνή φόρα να μας ακολουθήσουν. Και για εκείνες τις χώρες οι οποίες καθυστερούν και δεν δείχνουν διατεθειμένες να καταπολεμήσουν την φοροαποφυγή, έχουμε προτείνει την υιοθέτηση μιας μαύρης λίστας και την υιοθέτηση κυρώσεων. Κάτι άλλο που μας δείχνουν τα Panama Papers είναι ότι παραμένουν κενά και παραθυράκια στο νομικό πλαίσιο, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να τα κλείσουμε, εάν θέλουμε να επιτύχουμε την καταπολέμηση της ε, φοροαποφυγής. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με άλλους διεθνείς οργανισμούς και διακρατικούς οργανισμούς ε, του ΝΟΣΑ, των G, τους G20 και θα ήθελα να τονίσω τη μεγάλη ε, συνεισφορά που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να ε, παραμένει η δυναμική, η πολιτική δυναμική ισχυρή. Οι Υπουργοί Οικονομικών συναντήθηκαν πρόσφατα, θα συζητήσουν μάλλον, ε, πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Και από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει ε, συγκεκριμένα βήματα και ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Και τώρα έρχομαι σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχουμε διαπιστώσει ότι με ευφυεί ευφυείς δράσεις στοχευμένες και με πολιτική βούληση καταφέρνουμε να έχουμε αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσπαθήσει να ανταποκριθεί με συνολικό τρόπο, με ολιστικό τρόπο, στο δημόσιο αίτημα να είναι δικαιότερη η ε, φορολόγηση. Πρώτα απ' όλα, να υπάρχει διαφάνεια μεταξύ κρατών μελών με την ανταλλαγή των πληροφοριών ε, μέσω των εκθέσεων αναχώρα που αφορούν στις ε, συμφωνίες τύπου tax rulings. Και ε, πρόσφατα επεκτάθηκε το σύστημα αυτό, έγινε ακόμα διαφανέστερο. Μιας και υιοθετήσαμε μία από τις, ένα από τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καταστήσαμε τις πληροφορίες αυτές δημόσια διαθέσιμες. Προσπαθούμε λοιπόν να καταπολεμήσουμε αυτή τη διάβρωση της φορολογικής βάσης, τη μετατόπιση των κερδών, την δημιουργία σχημάτων όπως αυτά που διαπιστώσαμε μέσω των εγγράφων του Παναμά. Επίσης, τονίζουμε τη σημασία που έχουν ε, μέτρα όπως τα προτιμησιακά καθεστώτα. Συνολικά, όλα αυτά τα μέτρα θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον καλύτερο και για τις επιχειρήσεις και δικαιότερο και για τους πολίτες ε, εντός της Ένωσης. Έχουμε τρεις κυρίους στόχους. Πρώτα απ' όλα να υπάρχει ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο να διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε επιχείρηση δραστηριοποιείται εντό του έδαφου τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώνει ε, δίκαια το φορολογικό βάρο που τη αναλογεί εκεί όπου έχει ε, δημιουργήσετε τα κέρδη της. Ε, βεβαίως δεν μιλούμε για ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές. Αυτά είναι εθνικές αρμοδιότητες και ε, σεβόμαστε την αρχή της επικουρικότητας. Ωστόσο, οι αποφάσεις των κρατών μελών για τους φορολογικούς συντελεστές θα πρέπει να λαμβάνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην δημιουργείται ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών και να μην πρέπει κάποιο κράτος να αντιμετωπίσει τις διπλωνές επιπτώσεις άλλων αποφάσεων. αυτή τη στιγμή. Κάποια κρατημέλη αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να προστατεύσουν τη φορολογική τους βάση και να καταπολεμήσουν τη φοροαποφυγή, αλλά δυστυχώς υπονομεύονται αυτές οι προσπάθειες τους εξαιτία αποφάσεων των γειτόνων τους. Επίσης, επιχειρήσεις ε, εθνικές έχουν να αντιμετωπίσουν πολυεθνικές οι ε, είναι πρωταθλητές στην φοροαποφυγή. Έχουμε υπολογίσει ότι οι εθνικές ε, επιχειρήσεις επιβαρύνονται κατά 30% περισσότερο από τις πολυεθνικές. Εάν λοιπόν θέλουμε να δημιουργήσουμε ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού, θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των φορολογικών πολιτικών. Το ίδιο ισχύει και για το εταιρικό δίκαιο, στο, το οποίο είναι πεπαλαιωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί ε, προβλήματα άνευ λόγου στις επιχειρήσεις που θέλουν να διαδραστηριοποιούν ε, διασυνοριακά. Οι επιχειρήσεις επιθυμούν σταθερότητα. Είναι το σημαντικότερο για να είναι μια οικονομία ανταγωνιστική. Και ο μόνος τρόπος να το επιτύχουμε αυτό είναι να υπάρξει μια συνεκτική πολιτική συντονισμού των φορολογικών αποφάσεων, των φορολογικών πολιτικών. Τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει ε, υποχρεώσεις στο πλαίσιο του UBEPS, της ε, πρωτοβουλίας τη διάφορας της βάσης και της ε, μετατόπισης των κερδών και έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν σχετικά μέτρα. Αυτό θα πρέπει να γίνει γρήγορα, αλλά δεν υπάρχει λόγο να θεωρούμε ότι το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να βρει μόνο του τη λύση και να εξειδικεύσει την πρωτοβουλία BEPS ξεχωριστά. Γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα καταλήξουμε σε 28 διαφορετικές ε, νομοθεσίες οι οποίες θα δημιουργήσουν ακόμα περισσότερα προβλήματα στις επιχειρήσεις εξαιτία των διαφορών μεταξύ τους. Εμείς προσπαθούμε με πολλές ε, πρωτοβουλίες και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και με τα, εθνικά, και, και με τα κράτη-μέλη να το προλάβουμε αυτό. Επαναλαμβάνω ότι σεβόμαστε πλήρως την εθνική κυριαρχία. Το γεγονό ότι αυτές οι αποφάσεις είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Προσέχουμε πάντα να τηρείται η αρχή της επικοροτικότητα και της αναλογικότητας. Και επιδιώκουμε να υιοθετούμε πάντα το προσφορότερο νομικό μέσο. Ορισμένες, σε ορισμένες περιπτώσεις όταν ε, το ζήτημα είναι ε, ξεκάθαρα διασυνοριακό ή όταν αφορά πλήρως την ενιαία αγορά, μπορεί να χρειάζεται υιοθέτηση κανονισμών. Κάτι τέτοιο συμβαίνει, για παράδειγμα, στι προτάσει που υποβάλαμε τον Ιανουάριο. Εδώ χρειάζεται μια δεσυνοριακή προσέγγιση. Σε άλλε περιπτώσει, δίνουμε μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τις αποφάσεις τι δικές τους εθνικές συνθήκες, όπως ε, ε, για παράδειγμα κάναμε στον τομέα των διμερών συμφωνιών ε, αποφυγής διπλής φορολόγησης. το 2015 για παράδειγμα, εθελοντικά τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν στην, α, στην πρόταση, στην πολιτική που αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα δίνονται φοροαπαλλαγές για την έρευνα και την ανάπτυξη της επιχειρήσης. Μετά από, σε, ένα τέτοιο θέμα λοιπόν η εθελοντική ε, δέσμευση που συνοδεύεται και από μια αξιολόγηση μεταξύ κρατών μελών, λειτουργεί καλά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει και άλλες πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα τη CCCTV, για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιριών. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει προτάσεις αλλά για να αρχίσουν να υλοποιούνται χρειάζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Και γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί έχει υποστηρίξει θεναρά την υιοθέτηση πολιτικών στο θέμα αυτό. Το ίδιο και τα εθνικά κοινοβούλια. Ας το αξιοποιήσουμε αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο και ας αξιοποιήσουμε ως τον περισσότερο τον πολιτικό διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Με το κύρος που έχουν τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να πιέσουν τις κυβερνήσεις να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Και σε αυτό το πλαίσιο υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε είναι διατεθειμένη και με χαρά δέχεται τις προτάσεις ε, και ε, τις παρατηρήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Λαμασού για την διοργάνωση της σημερινής ε, συνάντησης και για την πρόσκληση. ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθυντά. Ας περάσουμε τώρα στην φάση της ανταλλαγής απόψεων. Μετά από τους παρόντες τέσσερις Προέδρους Επιτροπών, θα δώσω το λόγο σε όσους τον ζητούν. Παρακαλώ, κάντε την αίτηση γραπτός. Έχετε λάβει έντυπα. Και θα δώσουμε ανά δύο ε, εκπροσώπους εθνικών βουλών και πρώτα ο κύριος Χρήστος Γιάλας, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής των Πέντε λεπτά παρακαλώ. Κύριε Βιάλα. Ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ε, συζητάμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όλες τις ε, κοινωνίες, σε όλα τα κράτη-μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όλου του κόσμου. Ε, η φοροδιαφυγή και το χρήμα το πώς αυτό διαχέεται σε όλο τον κόσμο το οποίο φόρα αποφεύγει, δημιουργεί πλούτο αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία που είναι ο του ανταγωνισμός. Γιατί ποιος ο λόγος κάποιος να έχει ποσοστά κέρδους όταν μπορεί και φοροκλέπτει τους έμεσους φόρους αλλά ταυτόχρονα φοροαποφεύγει και τους άμεσους φόρους. Ενώ έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δημιούργησε την Νομισματική και Οικονομική Ένωση. Παρ' όλα αυτά, 16 χρόνια μετά, έχουμε μόνο Νομισματική Ένωση και η Οικονομική της Ένωση μένει αρκετά πίσω. Πιστεύω ότι με την ευκαιρία όλων αυτών των οποίων βγήκαν στο φως δημοσιότητας, όσον αφορά με τα Panama Papers και τις τεράστιες φοροδαφυγές που υπάρχουν, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αρχίσουμε να συζητάμε ε, σοβαρά και να το θέτουμε στη βάση του ακόμη και για ενιαίους συντελεστέ τουλάχιστον στους έμεσους φόρους, ειδικά των εμπορευμάτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών. Θα έλεγα ότι η έμεση φόρη, ο φόρος έμεσες αξίας θα ε, πρέπει να έχει μια ενοποίηση ή τουλάχιστον κατώτερους συντελεστές και ανώτερους για να σταματήσει και αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τους φορολογικούς παραδείσους, οι οποίοι είναι σε δύο, σε δύο επίπεδα. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός. Όμως όλη αυτή η φορολογική παράδειση δημιουργούν τον αθέμητο ανταγωνισμό, δίνουν, α, δημιουργούν τεράστια προβλήματα σε χώρες οι οποίες έχουν υψηλό ποσοστό, υψηλό ποσοστό φοροδιαφυγής και μία από αυτές τις χώρες είναι και η χώρα μας, στην οποία όμως δεν τις δίνουν και τη δυνατότητα οι γειτονικέ χώρε, οι οποίε έχουν πολύ χαμηλότερου συντελεστέ και λειτουργούν ω φορολογική παράδειση, να μπορέσει να αναπτυχθεί και ταυτόχρονα να βγει από την κρίση την οποία έχει περιέλθει ε, όπω ε, συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Όμω όλο αυτό το κύκλωμα τη φοροαποφυγή και τη διακίνηση του χρήματο, του μαύρου χρήματο, δεν γίνεται από μόνο του. Γίνεται βοήθεια τραπεζών. Άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη ότι θα θέσει κανόνες οι οποίοι θα θέτουν ε, τέρμα σε, σε αυτά τα κανάλια της φοροδιαφυγής και της κίνησης του μαύρου χρήματος. Πιστεύω ότι ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχει κοινά χαρακτηριστικά για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε μια εναρμόνιση φορολογικών ε, πολιτικών και να μπορέσουμε πραγματικά να θέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο το οποίο το οραματίστηκαν οι ευρωπαϊστές και οι γεννήτωρες αυτής, αυτού του μεγάλου εγχείρηματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται άμεση και πιστεύω ότι ειδικά στην λειτουργία των εταιριών εντός της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορεί να λειτουργεί μια ενιαία βάση δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι με την έναρξη εργασιών της κάθε εταιρεία μέσα από τη διασύνδεση των φορολογικών αρχών των κρατών μελών θα πρέπει να υπάρχει σε ενιαία βάση δεδομένων οπότε αυτόματα να γίνεται και ανταλλαγή των πληροφοριών όσον αφορά για τις δραστηριότητε των εταιρεών αυτών εντός των χωρών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νομισματική, οικονομική και νομισματική ενοποίηση της, της Ευρώπης δεν μπορεί να έρθει με όλη αυτή την διαφορετική αντιμετώπιση των εταιριών και των επιχειρήσεων. Θα πρέπει και σε δεύτερη φάση, ακόμη και, στους, ε, και στα ποσοστά και στους φορολογικούς συντελεστές των ποσοστών των άμεσων φόρων, να υπάρξει μίνιμουμ και μάξιμουμ ποσοστό φορολόγησης για να μπορεί έτσι κάθε χώρα να δημιουργεί το δικό της, α, τις δικές της πολιτικές εντός των ορίων. Όμως έτσι θα έχουμε δώσει το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ενιαία και έρχεται απέναντι σε, όλες, σε όλη τη διακίνηση αυτού του μαύρου χρήματος. Ελπίζω να είναι σημαντικές οι αποφάσεις, να μην μένουν μόνο στην διαδικασία των οδηγιών, αλλά να παρθούν στο επόμενο διάστημα και γρήγορα άμεσα και να είναι δεσμευτικές από όλες τις χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακολουθεί ο Πρόεδρος Μάσιμο Μουκέτη, Πρόεδρος της Επιτροπής για Βιομηχανία και Τουρισμό της Ιταλικής Γερουσίας. Επίσης πέντε λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες και αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι. Με την κοινοποίηση της 28ης Ιανουαρίου 2016 προς Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να προβεί στα απαραίτητα διαβήματα για να ανακόψει την επιθετική φορολογική πολιτική των εταιριών, τα γνωστά tax ruling, και να αποκαταστήσει την ελεύθερη, τον ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ των φορολογικών συστημάτων. Όμως, οι νομοθεσίες μας είναι απειθιωμένες Και αυτό αποδείχνεται από τον τρόπο που ορίζονται οι φόροι των επιχειρήσεων. Να μην λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μονομερή μέτρα. Δεν το, δεν το δεχόμαστε αυτό. Γιατί υπάρχει λόγος. Και σχετικά με τις μελλοντικέ συναντήσεις με Αμερικανούς εκπροσώπους, αλλά και στη συνεργασία με τον ΟΣΑ, όπως αναφέρει και ο πρόεδρος Λαμασού, προβλέπεται αυτή η συνεργασία, Όμω, οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενδέχεται να επιτρέψουν στις εθνικές κυβερνήσεις ε, να ε, ξεφύγουν από τις υποχρεώσει τους. Πρόκειται για κάλυψη. Κομψή μεν, αλλά όχι αποτελεσματική. Δεν μπορεί κανείς να αποφύγει εν τέλει ε, νομίζω εν υπάρχει ένα παράδειγμα από την Ιταλία. Ε, Ιταλικά δικαστήρια προέβησαν σε έρευνες κατά Google, Facebook και άλλων μεγάλων πολυεθνικών ομίλων σχετικά με, και μάλιστα με ενίσχυση των αρμοδίτων των φορολογικών αρχών. Εδώ πρόκειται για αρκετά εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα συμμετέχουν και ορισμένες ε, ε, μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, ε, θίγονται και μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πάει τώρα η Ιταλική δικαιοσύνη να υποκαταστήσει εξ ανάγκης την ε, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Και οι αποφάσεις οι οποίες είναι χρήσιμες δεν λαμβάνονται ωστόσο εν τέλει ή λαμβάνονται με προβολικά μεγάλη καθυστέρηση. Τι απαντά η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λέγει ότι γίνεται ε, προσπάθεια Η έδρα της επιχείρησης είναι μια έννοια αόριστη. Για, ξεκινά μάλιστα από το 19ο αιώνα. Έχει για πολύ καιρό καλύψει παράνομες δραστηριότητες. Όμως, κινδυνεύουμε να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στην πραγματικότητα των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Δεν έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να εντοπίσουμε την φορολογική βάση. Οι πολυεθνικοί αυτοί όμιλοι ακολουθούν μια επιθετική φορολογική πολιτική. Επιλέγουν τις χώρες τις οποίες θα δηλώσουν τα κέρδη τους. Ανάλογα με τους βολεύει. Και τελικώς το ρευστό καταλήγει σε φορολογικούς παραδείσους. Ορισμένες ε, χώρες έχουν επιτύχει να προσελκύσουν με χαμηλού φορολογικού συντελεστές τι μεγάλε πολυεθνικέ επιχειρήσει, αυτό όμως ζημιώνει τις άλλες. Εν τέλει αυτό που λείπει είναι η ασφάλεια. Και αυτό επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο και δεν αρκούν οι προσπάθειες της δικαιοσύνης. Η Ιταλική Γερουσία σύστησε στην κυβέρνηση να εξετάσει εάν δεν έχει έρθει η ώρα πράγματι να δηλώνονται επιγραμμικά, online δηλαδή, οι δραστηριότητες των Ιταλικών επιχειρήσεων και αυτές που έχουν σχέση με το εξωτερικό. Όμως ή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορολογικός αριθμός και θα υπάρχει μετά μία έδρα με βάση τον αριθμό αυτό και επομένως θα εκδίδονται ισολογισμοί που θα είναι δυνατόν να ελεγχθούν ή θα επιβάλλεται μια φορολογία στα εισοδήματα της επιχείρησης σε ένα ορισμένο συντελεστή που θα επιβάλλονται και στις θηγατρικές επιχειρήσεις. Πάντως η Ιταλία δεν πρόκειται να αναλάβει με ονομερός ενέργειες. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει τώρα ο πρόεδρος Ερικ Μπάνκι, που είναι πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Ουγγρικής Βουλής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής της Ουγγρικής Βουλής να σε ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να έρθουμε και να συζητήσουμε μαζί σας και με εκπροσώπους ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων των Ευρωπαϊκών χωρών. Θεωρούμε το θέμα της φοροαποφυγής και η πάταξη, η αντιμετώπιση της φοροαποφυγής είναι πολύ σημαντικά θέματα. Και μία σημαντική αλλαγή και πρόκληση και για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Οι πολυεθνικές εταιρείες και όμιλοι χρησιμοποιούν περίεργες φορολογικές δομές και μετατοπίζουν τα κέρδη τους ε, από την χώρα που πραγματοποιούν τις δραστηριότητές τους και παράγουν τα κέρδη τους. Το πιο σημαντικό πάντως είναι να προσπαθήσουμε να ε, καταπολεμήσουμε αυτή την απώλεια φορολογικών εσόδων και να φορολογούμε τις εταιρείες εκεί που πραγματοποιούν τα κέρδη και δημιουργούν αξία. Για παράδειγμα, στην Ουγγαρία Είχαμε πρόβλημα με τα φορολογικά έσοδα, κυρίως γιατί είχαμε εταιρείε ε, με πολλές έδρες. Και έτσι χρησιμοποιούσαν προνομιακά φορολογικά καθεστώτα για να καταβάλουν το χαμηλότερο δυνατό φόρο. Καταφέραμε να θέσουμε ένα τέρμα στην πρακτική αυτή των ε, επιχειρήσεων. Και φορολογήσαμε τις επιχειρήσεις εκεί που ε, παρήγαν αξία και κέρδη. με βάση δηλαδή την ε, συντάξη που ίσχυε στη συγκεκριμένη περιοχή. Θεωρούμε ότι και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει οι φορολογικές διατάξεις να εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Όπως είπαν όμως και οι συνάδελφοι από την Ιταλία και την Ολλανδία, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πρόσφορο και ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον που δεν θα αναγκάζει τις εταιρείες να μετατοπίσουν τα κέρδη τους. Και έχουμε ένα φορολογικό συντελεστή 19% για τις επιχειρήσεις. Θεωρούμε ότι έτσι δημιουργείται ένα ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον. Είναι σημαντική και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων για να γίνει αποτελεσματική η διαδικασία και θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταλλαγή των πληροφοριών. Ο Ιταλός συνάδελφος μίλησε για τις ε, πολυεθνικές ε, εταιρείε που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και πώ θα πρέπει να φορολογούνται, μια και τιμολογούν μέσω διαδικτύου τα αγαθά του. Και είναι πολύ δύσκολο ο έλεγχο ε, των κινήσεων τη παροχή υπηρεσιών και αγαθών. Και αυτό είναι και δύσκολο να φορολογηθούν αυτέ οι εταιρείε του διαδικτύου δεν ξέρουμε ακριβώς πού παράγουν τα κέρδη τους. Η Ουγγαρία είναι υπέρ του συντονισμού με τις υπόλοιπες χώρες μέλη και με τις ε, χώρες όσα. Και θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα αγαστό περιβάλλον συνεργασίας και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Βέβαια, θα πρέπει να διαφυλαχθούν και οι εθνικές αρμοδιότητες στα θέματα αυτά. Η Ουγγρική κυβέρνηση και η Ουγγρική Βουλή προσπαθούν να εξετάσουν τους κανόνες και να τους αναθεωρήσουν εν ανάγκη για να αποκαταστήσουν αποτελεσματικά φορολογικά μέτρα. Θα χρειαστούμε και νέες νομοθετικέ διατάξεις για να διαμορφώσουμε ένα περίπλοκο αλλά ενοποιημένο νομικό περιβάλλον για να αντιμετωπίσουμε τη φοροαποφυγή. Στην Ουγγαρία και η κυβέρνηση και η Βουλή περιμένουν τέτοιες ευρωπαϊκές προτάσεις για να τις μεταφέρουμε και στην εθνική μας ένωμη τάξη. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι τέτοιου είδους συνεργασία δεν μπορεί να αντιβαίνει να σφετερίζεται τις εθνικές αρμοδιότητες για τη φορολογία. Χρειάζεται όμως οπωσδήποτε μια διαφάνεια και μάλιστα ενισχυμένη. Γι' αυτό εμείς έχουμε ένα σύστημα ταμιακών μηχανών online και έτσι μπορούμε να ελέγχουμε τα φορολογικέ τις φορολογικές κινήσεις με πολύ καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ και καλή τύχη εύχομαι σε όλους μας. Σας ευχαριστώ. Τέλος θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Ξέγκος Μπιερέτσκι, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού και Δημοσίων Οικονομικών της Πολωνικής Γερουσίας. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω κύριε Λαμασούρ για την οργάνωση αυτής της ε, συνάντησης και να ευχαριστήσω και την Ολλανδική Προεδρία για την άσκηση πίεσης προκειμένου να ε, λυθεί το πρόβλημα αυτό το συντομότερο δυνατό. Οι πολυεθνικές εταιρείες και όμιλοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση και τις αναντιστικές των φορολογικών συστημάτων για να φοροαποφύγουν τις υποχρεώσεις τους. Και αυτό πραγματικά μας ε, ε, εκνευρίζει και μας ενοχλεί ιδιαίτερα στην Πολωνία. Μάλιστα κάποιες ε, τερά... μεγάλες πολυεθνικές ε, καταβάλουν ε, συμβολικούς και μηδενικούς φόρους. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα που μας εξοργίζει ιδιαίτερα και αποτέλεσε και σημαντικό σημείο στην προεκλογική μας εκστρατεία και μάλιστα μας έδωσε την νίκη στις εκλογές. Η αύξηση των κερδών των μεγάλων πολυεθνικών ομιλών δεν έχει αντίκρισμα σε αντίστοιχη κοινωνική ευημερία και ανάπτυξη. Γι' αυτό και θα πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να αποκαταστήσει μεγαλύτερη δικαιοσύνη και ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα φορολογίας των νομικών προσώπων και των εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την αποτελεσματικότητα των αλλαγών αυτών και των νέων μέτρων ε, θα εξαρτηθεί και η περαιτέρω συνεργασία μας. Ή μάλλον, ε, η η συνεργασια μας είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων. Ε, με τέτοια αποτελέσματα θα έχουμε μια δίκη φορολόγηση των εταιριών στις χώρες που πραγματικά έχουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες και που παράγουν τα κέρδη και την οικονομική τους αξία. Θα πρέπει να φορολογούνται εκεί που παράγουν τα κέρδη, τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις μερικές από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και θα επηρεάσουν ιδιαίτερα την οικονομία πολλών χωρών και γι' αυτό θα είναι δύσκολο πιστεύω να τεθούν σε εφαρμογή σχετικά γρήγορα. Για παράδειγμα το CCCTB, η Κοινή Ενωπημένη Βάση Φορολογίας Εταιριών. Ε, δεν νομίζω ότι θα εφαρμοστεί γρήγορα. Ε, θα πρέπει όμως ε, να ε, εγκρίνουμε όλες τις προτάσεις που στόχο την βαθμιαία προοδευτική εφαρμογή της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιριών. Επίσης, το, η υποχρεωτικότητα του συστήματος ε, για τις πολυεθνικές κυρίως εταιρείε. Ένα τέτοιο υποχρεωτικό χαρακτήρα δεν μπορεί να γίνει αυτόματα δεκτό. Θα πρέπει να συνοδευτεί από ανάλυση διεξοδική πολύ πιο ε, συγκεκριμένων προτάσεων. Επίσης, ε, είμαστε κατά μιας λύσης που θα μπορούσε να περιορίσει ή να κλονίσει την ε, ε, κατοχυρωμένη στη συνθήκη ελευθερία παροχής υπηρεσιών. αναφέρθηκε το θέμα της εναρμόνισης της άμεσης φορολογίας από ένα προλαλήσαντα. Τα κράτη-μέλη όμως ε, αυτόνομα ε, καθόρισαν την πολιτική τους για την έμεση φορολογία. Και δύσκολο θα είναι η εφαρμογή υποχρεωτικών διατάξεων στην περίπτωση αυτή. Μόνο συστάσεις μπορούν να γίνουν δεκτές. Επίσης, με ικανοποίηση ε, δέχομαι την ε, νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, φυσικά θα πρέπει να συγκεκριμενομηθούν αυτές οι προτάσεις και ίσως να διαγραφούν ή να βληθούν κάποιες πιο αυστηρές διατυπώσεις, αλλά κάτι τέτοιο προϋποθέτει μια πιο συστηματική ανάλυση. Πάντως, σίγουρα στην Πολωνία θα χρειαστούμε πολύ περισσότερο χρόνο για να προβούμε σε πιο εμβριθή ανάλυση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Πολωνία αναγνωρίζει τη σημαντική αλλαγή της οδηγίας για τα θέματα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και το θέμα του country by country reporting, των εκθέσεων αναχώρα. Πάντως είναι, θετική η κατέθεση των δράσεων και των μέτρων που προτείνονται στη σχετική αναθεώρηση της οδηγίας. Γενικώ η γερουσία της Πολωνίας θεωρεί ότι ο στόχος ε, της πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αξιέπαινος και χρήζει αμέριστης υποστήριξης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στρέφουμε προς τους δύο συνεισηγητές. Για δύο λεπτά ο καθένας σας για να αναπτύξετε λίγο τι αναμένετε από την ε, παρούσα συνάντηση. Γέπε Κόφοντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πρώτα πρώτα ευχαριστώ ως συνεισηγητής όλα τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που διέδεσαν τον χρόνο τους για να προσέλθουν εδώ. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι είναι ενδιαφέρον διότι έχουμε ενώπιό μας ένα θέμα το οποίο είναι εθνικής αρμοδιότητας. Η συλλογή, δηλαδή η των φόρων. Έχουμε όμως από τη μια μεριά και μια παγκόσμια διάσταση. Βλέπουμε δηλαδή ότι παρόλο που είναι εθνική αρμοδιότητα, καμιά φορά είναι δύσκολο να εκπληρωθεί αυτή η εθνική αρμοδιότητα, διότι υπάρχουν αυτοί που φόρο αποφεύγουν και φόρο διαφεύγουν και ανά τον κόσμο. Είδαμε και την ιστορία αυτή με τα έγγραφα του Παναμά. Ποιο είναι ο κοινό μα στόχο, ημών δηλαδή και εθνικών και ευρωπαίων βουλευτών, ότι θα διαθέτουν δηλαδή οι εθνικέ βουλέ την πραγματική εξουσία να εισπράττουν φόρους και από την άλλη μεριά να εξασφαλίσουμε φορολογική δικαιοσύνη και για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες. Διότι αυτό που συμβαίνει τώρα το εξήγησε και ο πρόσωπος της Κομισιόν. Αν δείτε για παράδειγμα την φορολογική επιβάρυνση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι 30% παραπάνω από τις μεγάλες πολυεθνικές. Αυτό σημαίνει αθέμητο ανταγωνισμό που βαρύνει μεγάλο μέρος της κοινωνία μας, δηλαδή των μικρών και μεσών επιχειρήσεων, που είναι εκείνε οι οποίες δημιουργούν απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου μιλήσαμε και για τα γνωστά Panama Papers, που δεν είναι βέβαια αρμοδιότητας της Επιτροπής Τάξε, της δικής μας εδώ Επιτροπής, αλλά γνωρίζουμε όμως ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι η διαφάνεια, η συνεργασία με τι άλλε χώρε και με τι άλλε δικαιοδοσίε απανταχού του κόσμου. Και ιδίω χρειαζόμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ισχυρό παίκτη στο πεδίο αυτό και τα όσα αποφασίζει να φροντίσει να προβληθούν και να εφαρμοστούν και παγκόσμια. Έχω βέβαια μόνο δύο λεπτά, αλλά θεωρώ ότι έχουμε μια κοινή ατζέντα που όλοι πρέπει να εγγύψουμε σε αυτήν ο καθένας από την σκοπιά του, από τη γωνιά του. Ως συνεισηγητή λοιπόν, αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον όλες τις προτάσεις, συστάσει και ιδέε σα. Ευχαριστώ κύριε εισηγητά. Ο άλλο συνεισηγητή τώρα, ο κύριο Μιχαήλ Τόερελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ και αγαπητοί συνάδελφοι των Εθνικών Κοινοβουλίων, θα ήθελα πρώτα να τονίσω πόσο σημαντική είναι η παρουσία σας σήμερα εδώ, 19 χώρες μέλη. Είναι σπουδαίο αυτό για μας. Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι μόνο με κοινή προσπάθεια. Ως συνηγητής των δύο επιτροπών για τα φορολογικά, είναι, θεωρώ ότι είναι σημαντικά τα συμπεράσματα των επιτροπών μας, των εργασιών της Επιτροπής μας. Πρόκειται για ε, μια προσπάθεια συντονισμού 28 ιδιαίτερα περίπλοκων φορολογικών συστημάτων για την αποκάλυψη των παράθυρων που ε, έχουν μέχρι τώρα εκμεταλλευτεί οι διεθνεί και πολυεθνικές ιδίω επιχειρήσεις. Αν θέλουμε να ανακόψουμε την πορεία αυτή χρειαζόμαστε μια κοινή αγορά όπου η ελευθερία της διακίνησης των κεφαλαίων θα ακολουθεί, θα σέβεται κάποιου κοινού κανόνες. Γι' αυτό και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ψηφίσει νομοθεσία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, για παράδειγμα, επίσης για την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση εταιριών, για να μην γίνεται ο ανταγωνισμός στην βάση της διάβρωσης φορολογικής βάσης και μετατόπισης κερδών, αλλά μόνο στη βάση των συντελεστών. Και τότε θα μείνει μόνο η εξωτερική διάσταση. Την εξωτερική διάσταση αυτή μας έχει μείνει ένα είδος υπόλοιπο γιατί έχουμε και όλη την ιστορία των φορολογικών παραδείσων, τις απαγορεύσεις διπλών φορολογήσεων. Αυτά βέβαια έχουν πει σε μια διαδικασία διερεύνηση σε σχέση με τα έγγραφα του Παναμά και τουλάχιστον κάθε κέρδος το οποίο φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τουλάχιστον άπαξ, μια φορά δηλαδή φορολογηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κάποιο σύστημα, το οποίο θα συζητηθεί βέβαια. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις σας και την συζήτηση και εύχομαι να μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό τρόπο να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο BEPS, διότι θεωρώ ότι όλων το συμφέρον τελικώς υποσκάπτεται εφόσον υπάρχει αυτή η επιθετική φορολογική πολιτική. Ωραία. Περνάμε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων. Όπως είπα θα δίνω το λόγο πρώτα σε δύο βουλευτές και μετά σε έναν ευρωβουλευτή. Θα με αυτούς που έστειλαν και γραπτό στις ε, παρατηρήσεις τους από την Βουλή των Κοινοτήτων. Ε, σας ευχαριστούμε θερμά. Μας τιμά ιδιαίτερα, Λόρα Ντέιβις, η παρουσία εδώ. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ολλανδική Προεδρία για την ευκαιρία που μας δώσατε να λάβουμε μέρος στη συζήτηση. Θα ξεκινήσω με μερικά σχόλια που ίσως φανούν αρνητικά, αλλά ε, ίσως ε, σας βοηθήσουν και στο τέλος θα κάνω και ένα θετικό σχόλιο. Νομίζω ότι υπάρχει μια σύγχυση στην ορολογία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πολλές φορές αναφέρεται ε, η αφοροαποφυγή και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός. Ε, ε, ε, είναι, ε, δεν είναι ταυτολογία γιατί εναλλακτικά χρησιμοποιούνται. Υπάρχει όμως διαφορά μεταξύ τους. Ε, και στις δύο περιπτώσεις έχουμε νόημα πράγματα. Ένα, η φόρο διαφυγή, η tax evasion είναι αξιόπινη πράξη. Αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ φόρο αποφυγής αφενός και φόρο διαφυγής αφετέρου και φορολογικού, επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού θα πρέπει να διευκρινίσουμε το περιεχόμενο έννοιας, γιατί η σύγχυση αυτή στην ορολογία μεταφράζει και μία σύγχυση στην πράξη. Σε έναν ιδεώδη κόσμο, ίσως ε, θα έπρεπε η φορολογία να είναι κοινοτική αρμοδιότητα. Όπω όμω μα υπενθύμησαν οι συνάδελφοι, ε, η φορολογία δεν αποτελεί κοινοτική αρμοδιότητα, αλλά εθνική αρμοδιότητα. Και είναι και επικίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να επιλύσει ένα πρόβλημα που δεν είναι σε θέση να το κάνει. Γιατί έτσι ίσω γύρει προσδοκίε που δυστυχώ διαψευθούν και οδηγήσουν μεγάλη ματέωση και απογοήτευση. Και δεν μπορεί να γίνει ε, κάτι ε, για την φοροαποφυγή, να μετατραπεί αυτή σε αξιόπινη πράξη, σε φοροδιαφυγή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά μόνο σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, με την ιδιοθέτηση ενός γενικού κανόνα φοροαποφυγής, ε, που το έχουμε ε, τελευταία εφαρμόσει στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι θετικό, γιατί για πολλά χρόνια μας ξεγελούσαν επιχειρήσεις μεγάλες όπως η Google και η Starbucks. Έτσι, μία εμπορική συναλλαγή μπορεί να θεωρείται τεχνική και μόνο για λόγους φορολογική απαλλαγής. Σε τέτοια περίπτωση ε, εισπράτε παρόλα αυτά φόρους να μην υπήρχε προηγούμενη συμφωνία. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά των κρατών μελών που είναι και αρμόδια για τη φορολογική πολιτική. Τώρα, το θετικό σχόλιο. Με προβληματίζει η θέση που έχει λάβει η Επιτροπή για τι φορολογικέ ευθύνε. Βέβαια, θα πρέπει να αναλαμβάνονται ευθύνε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποκαθίσταται η διαφάνεια στον τομέα αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τι οδηγίε, Να, ε, να προτείνουν τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών αλλά υπάρχει και εδώ μια σύγχυση στα χαρτιά, για παράδειγμα. Στην πρώτη σελίδα, στην πρώτη παράγραφο, ε, εκεί ε, να υπάρχει ε, δημόσιος έλεγχος για το που καταβάλλεται ο φόρος και άρα να αποκαλύπτονται κάποια δημόσια έγγραφα. Ενώ πιο πέρα αναφέρεται ότι οι πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται στο κοινό. Υπάρχει μια σύγχυση. Στη μία αναφέρεται δημόσια πρόσβαση και στην άλλη αποκλείεται κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι δεν θα δίνονται πληροφορίες στο κοινό. Πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος, θα πρέπει να είναι δημόσια προσιτές αυτές οι πληροφορίες. Επίσης, ε, ε, ο περιορισμός στο, σε 750 εκατομμύρια τζίρο είναι υπερβολικά υψηλός. Νομίζω ότι όλες ε, οι εταιρείε, οι δημόσιες και ιδιαίτερα οι καταχωρισμένες στο χρηματιστήριο, καταχωρημένες στο χρηματιστήριο, συγγνώμη, στο χρηματιστήριο, έχουν ε, πολύ ε, ε, μεγαλύτερο τζίρο και νομίζω ότι και οι μέτοχοι αλλά και οι πελάτες έχουν δικαίωμα να, γνωρίζονται που καταβάλλονται, να γνωρίζουν που καταβάλλονται οι φόροι. Οπότε, αυτά για τις προτινόμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Είναι, παραλαμβάνει η φορολογία αθηνική αρμοδιότητα, αλλά σε θέματα αποκάλυψης πληροφοριών και διαφάνειας, εκεί θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο απαιτητικοί. Σας ευχαριστώ, Μιλόρδε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Πιέρα Λαμιουέ, που είναι αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής ε, Οικονομικών της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναγνωρίζω τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει στην Ευρώπη σε αυτή την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Αν σκεφτούμε πού ήμασταν πριν από τρία χρόνια, όταν οι G20 ξεκίνησαν αυτή την πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της διάβρωσης φορολογικής βάσης, ε, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι έχουμε ασχοληθεί με ένα θέμα δύσκολο στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι το ζητήματα αυτό είναι εθνικής ε, αρμοδιότητας, δηλαδή ε, αρμοδιότητα των εθνικών κοινοβουλίων. Αλλά με την δυνατότητα που έδωσε ο πρόεδρος Λαμασούρ να εμπλακούν και τα εθνικά κοινοβούλια, καταφέραμε να προχωρήσουμε γρήγορα και θα έλεγα ότι η πρωτοβουλία BEPS ήταν υποδειγματική για δύο λόγους. Πρώτον γιατί ε, δημιουργεί ισότιμο ανταγωνισμό εάν εφαρμοστεί σωστά, έναν ανταγωνισμό ο οποίος είναι απαραίτητος και δεύτερον γιατί γνωρίζουμε ότι στη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Επομένως, είναι απαράδεκτο να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή ο, ο ανταγωνισμός ε, μεταξύ ορισμένων κρατών ε, στον τομέα της φορολογίας ε, είναι απαράδεκτος. Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες πολυεθνικές ε, επιχειρήσεις καταφέρουν να πληρώνουν λιγότερους φόρους από τις μικρομεσαίες που έχουν έδρα σε μια χώρα μόνο. Λοιπόν, πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία, να υποστηρίξουμε ε, την πρόταση για τις εκθέσεις αναχώρα, που βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από άλλα κράτη του κόσμου, αλλά κατά την άποψή μου πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο από τις ε, ε πρωτοβουλίες του ΩΣΑ και να προχωρήσουμε στην εναρμόνιση των εταιρικών μορφών είναι ένα θέμα σημαντικό και για την κοινή αγορά και για την ΟΝΕ. Αυτή είναι η πιο θεμελιώδης, εάν θέλετε, ε, λύση για το, το πρόβλημα που θα δώσει την δυνατότητα μεγαλύτερης απλοποίησης του συστήματος, μεγαλύτερης διαφάνειας για τους πολίτες. Ένα θεμελιώδης λοιπόν μέτρο το οποίο μπορεί να το εξετάσει κατά την άποψή μου η Επιτροπή αυτή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην Ντανούτα Χούμπνερ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εσείς για δύο λεπτά. Δύο ή τρία. Τρία. Η κυρία Χούπνερ. Βεβαίως, τα τελευταία δύο χρόνια η κυρια χουμνερ βεβαιως τα τελευταια δυο χρονια η εργασια μας για την εταιρική φορολογία ε, έλαβε σημαντικές οθήσεις από πολύ δραματικά γεγονότα. Εάν εφαρμόσουμε τα όσα μας είπε ο ε, κύριος Quest, τα τρία αυτά πακέτα, θα πάμε και πάρα πέρα από την αντιμετώπιση των ε, επίκαιρων προκλήσεων και θα φτιάξουμε ένα σωστό φορολογικό σύστημα στην Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να είναι το καθήκον μας. Ένα θέμα που θέλω να θέσω εδώ και να πω λίγα λόγια σχετικά, έχει σχέση πάλι με αυτά που είπε ο Γενικός Διευθυντής κ. Quest, μια εξισορρόπηση μεταξύ λύσεων που είναι αναγκαίες για την εταιρική φορολογία στο εθνικό επίπεδο και από την άλλη μεριά των λύσεων που θα πρέπει να αρθούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο και βεβαίως και οι συστάσει του ΟΣΑ. Δηλαδή να βρεθεί μια σωστή ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που πρέπει να εγκριθούν και να γίνουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτά που πρέπει να γίνουν στο εθνικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όμω γενικά νομίζω ότι ω αποτέλεσμα θα έχουμε μάλλον ένα πλήθος νομικών εργαλείων και εργαλείων πολιτικής. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε εργαλεία πολιτικής σε διαφορετικά επίπεδα. Κάτι που σημαίνει επίσης ότι χρειαζόμαστε και ένα άνευ επίπεδο συνεργασίας και παρακολούθησης. Και έχω και το θέμα ότι η αντιμετώπιση των φορολογικών θεμάτων χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην δημοκρατική νομιμοποίηση πολύ περισσότερο μάλιστα στην, στις υποθέσεις της φορολογικής πολιτικής από τις άλλες πολιτικές. Εμείς καλούμεθα εδώ ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά βεβαίως και οι εθνικοί μας συνάδελφοι στο εθνικό επίπεδο, να προσφέρουμε την δημοκρατική νομιμοποίηση σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής για την διόρθωση του φορολογικού συστήματος, να γίνει δηλαδή δίκαιο αλλά και διαφανές και ασφαλές απέναντι σε οποιαδήποτε κατάχρηση. Αυτή η διπλή νομιμοποίηση με συμβολή και του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, και αυτό που χρειάζεται είναι η ενίσχυση πρώτα-πρώτα του πολιτικού διαλόγου. Και έρχομαι πάλι στον Στίβεν Κουέστ που ζήτησε συνεργασία. Χρειάζεται να ενισχύσουμε την συνεργασία. Όμως, τα Εθνικά Κοινοβούλια θα αναλάβουν και συγκεκριμένα την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΣΑ για να μεταμορφωθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι ευρωπαϊκές οδηγίες, καθώς και να παρακολουθούν την εφαρμογή τους. Αυτή η διαδικασία της διόρθωσης δηλαδή των φορολογικών συστημάτων στην Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό θα αναλυθεί ως ευθύνη από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτά θέλω να πω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Ντανούτα. Επανερχόμαστε σε εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβούλιων να δώσω το λόγο στον κύριο Πέντρο Σάουρα της ε, Ισπανικής Βουλής των Αντιπροσώπων. Τρία λεπτά κύριε Σάουρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά τη γνώμη μου, στον κόσμο που ζούμε έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγκόσμιες προκλήσεις και η φοροαποφυγή είναι μια τέτοια παγκόσμια πρόκληση και θα πρέπει να κάτσουμε όλες οι βουλές από κοινού και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κοινά προβλήματα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε, τα μέλη της Επιτροπής σας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί συμβάλλεται σε μια παγκόσμια αλλαγή του τρόπου σκέψης, ώστε να αποκαταστήσουμε μια πιο δίκαιη και πιο αξιοπρεπή φορολόγηση. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα ε, του, του τρόπου της διαμόρφωσης και της οργάνωσης κοινωνίας, αλλά ακριβώς αυτή η οικονομική κατάσταση ενέχει κάποιες ε, αδικίες και μπορούμε να τη διορθώσουμε με τη χρηματοδότηση του κράτους πρόνοιας και μιας κοινωνικής ευημερίας. Επίσης, ελπίζω ότι το έργο μας θα είναι καρποφόρο και ως προς το σκάνδαλο για τα έγγραφα του Παναμά, το Panama Papers και το Panama Papers. Έχουμε ένα επιπλέον βήμα για να προχωρήσουμε σε αυτή την παγκόσμια στρατηγική για τη φορολογία. Και στην Ισπανία ζητήσαμε μια εξεταστική επιτροπή για τη διαλεύκανση των εγγράφων του Παναμά. Και επίσης ε, θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε κάποια θέματα που κατά τη γνώμη μας είναι σημαντικά και σε αυτά θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε σαφή και σταθερή πρόοδο. Καταρχήν, το θέμα της κοινή ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιριών. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Θα πρέπει να το πραγματοποιήσουμε, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, γιατί είναι κατάλληλη στιγμή. Είχαμε πολλά χρόνια επιβράδυνσης αυτής τη πολιτική αυτού του φορολογικού μέτρου, αλλά τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να, δείξουμε και μεγαλύτερη φιλοδοξία από τον ΩΣΑ. Επίσης, ό,τι αφορά την, τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Φορολογικών Παραδείσων. Και αυτό είναι ένα βήμα πρόοδου και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την κατάλληλη στιγμή. Αυτή είναι η πρόσφορη στιγμή. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτό τον αγώνα δρόμου για τη φθηνότερη φορολογία. Γιατί κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο την ε, παγκόσμια κοινωνική συνοχή και την ε, Εθνική Κοινωνική Συνοχή. Επίσης το πρόγραμμα για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Καλό αυτό, αλλά θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι και να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος, ο ουσιαστικός δικαιούχος αυτών των συναλλαγών που αποκαλύπτονται χάρη σε αυτή την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε τελική ανάλυση πιστεύω ότι θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη φιλοδοξία γιατί και η στιγμή είναι κατάλληλη αλλά και το απαιτούν οι παγκόσμιες προκλήσεις και ο παγκόσμιος χαρακτήρας αυτών των προβλημάτων και προκλήσεων. Σας ευχαριστώ. Το τελευταίο σχόλιο που κάνατε είναι ένα συμπέρασμα που θα πρέπει να αντιλήσουμε από το θέμα των εγγράφων του, Καναδά, του Παναμά. Θα δώσω τώρα το λόγο και κάνω και στο συγγνώμη αν προφέρω Λάθο το όνομά σα. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Σλοβενίας, τον κύριο Τίλεμ Μπόζιτ. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ξεκινώντας να πω ότι η σλοβενική νομοθεσία φορολογική είναι αρκετά προηγμένη, αλλά βεβαίως πάντοτε είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για βελτίωση το Εθνικό μας Κοινοβούλιο έχει ε, βλέπει με θετικό μάτι με τέτοια, ένα τέτοιο ενδεχόμενο γιατί όλοι γνωρίζουμε τι κινδύνους ε, ενέχει η διάβρωση της φορολογικής βάσης. Η χώρα μου όπως και όλη η Ευρώπη ε, έχει πληγεί από την οικονομική κρίση επομένως έχει γίνει ακόμα σημαντικότερη η εισπράξη των φόρων. Τούτου λεχθέντος. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η συλλογή και η ανταλλαγή πληροφοριών. Ιδιαίτερα η συλλογή πληροφοριών εγκαίρως. Εάν λάβουμε υπόψη τον χρόνο που χρειάζεται για να φτάσουν μέχρι ε, στις φορολογικές αρχές οι πληροφορίες και να ε, τύχουν επεξεργασίας, ε, πολύ συχνά εκείνοι που είχαν εγκληματίσει έχουν φροντίσει να κρύψουν τα ίχνη τους και όλα είναι, φαίνονται τέλεια. Η ε, νομοθεσία της Σλοβενίας δίνει διάφορα εργαλεία ε, όπως η κοινοποίηση των φορολογικών συμφωνιών ε, και άλλα μοντέρνα εργαλεία, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς πώς δραστηριοποιούνται οι φορολογούμενοι. Αλλά το ερώτημα που εμένα με απασχολεί είναι μήπως δεν θα προλάβουμε να εξυγχρονίσουμε το σύστημα εγκαίρως η φορολογική παράδειση ε, υπάρχουν εδώ και 30 χρόνια. Και τώρα μόλις ξεκινούμε να τους ζητάμε και να εξετάζουμε τρόπους αντιμετώπισης τους. Ε, βεβαίως η πληροφορική μας δίνει κάποιες ε, λύσεις, αλλά μέχρι τώρα αυτό που αξιοποιεί το ήταν οι διαφορές στην εθνική νομοθεσία. Σήμερα βλέπουμε μια μετακίνηση προς ακόμα πιο εξελιγμένες τεχνικές, όπως για παράδειγμα οι ηλεκτρονικές πληρωμές με κρυπτογραφημένα νομίσματα στο ίντερνετ. Πρέπει λοιπόν να ε, βρισκόμαστε σε παγρύπνηση Προσπαθούμε να, να, να κάψουμε την οικονομική κρίση, αλλά αν καταφέρναμε να αντιμετωπίσουμε τη διάβνωση τη φορολογική βάση, καταφέρναμε φορολογική δικαιοσύνη, τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμα μεγαλύτερα. Σε... Χώρες όπως η Νιγηρία διαπιστώνουμε ότι τα φορολογικά έσοδα ε, είναι περίπου το 10% του, α, του, του εσόδων τους. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Σας ευχαριστούμε. Θα σημειώνω ότι ο Γενικός Διευθυντής της Αρμόδιας Διεύθυνσης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σημειώσει τις αντιρρήσεις, τις ανησυχίες που εκφράσατε, μάλλον για το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και το γεγονός ότι μπορεί να μην λειτουργεί τόσο γρήγορα. Επανερχόμαστε τώρα και θα δώσω στους ευρωβουλευτές και θα δώσω το λόγο στον Πίτερ Σάιμον από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πέτερ Σίμων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επανέρχομαι σε κάτι που είπε ο Γέπε Κόφοντ εκ των συνεισηγητών. Πρώτο, είναι θαυμάσιο που συναντώμεθα εδώ με βουλευτές των Εθνικών Βουλών που έχουν την κατεξοχήν αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά και όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα αυτό αποτελεί απόδειξη ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί πια καν να επιληθεί μόνο στο εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν όλοι πλέον. Όμως αν ξεκινήσουμε τώρα την πορεία αυτή ως συνολική Ευρώπη, και καλό είναι αυτό και θετικό και πολύ το είπαν μέχρι τώρα, είναι εξίσου σημαντικό κατά την άποψή μου να εξηγήσουμε όχι μόνο στους όμορους γειτονές μας, τα σχετικά με tax rulings, με την φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων, το reporting αναχώρα και ούτω καθεξής, είναι σημαντικό να τα εξηγήσουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Εξηγώ. Είδαμε στις διαδικασίες ε, διαφόρων ενισχύσεων. LuxLeaks, Amazon, πόσο σημαντικό είναι να έχουμε κάποιον ο οποίος, η οποία δηλαδή η Επιτροπή, είναι θεματοφύλακας των συνθήκων, δηλαδή στην ουσία το αστυνομικό όργανο που οφείλει να παρακολουθεί, να εξετάζει αν κάθε χώρα μέλος εξυπηρετεί, φροντίζει, τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες. Εάν στα πράγματα αυτά δεν είναι πλήρως ενήμεροι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε αφαιρούν οι χώρες μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δυνατότητα να ερευνήσει τις παραβίασεις αυτές και να τις διώξει. Και είναι πολλές οι χώρες μέλη αυτές. Είναι οι κυβερνήσεις σας. Πολλές από τις κυβερνήσεις σας που δεν το επιθυμούν. Σας παρακαλώ λοιπόν, με όλα αυτά που συζητούμε τώρα εδώ, με όλα αυτά που ερχόμαστε και λέμε οι μεν τους δε πόσο σημαντικά είναι. να ζητήσουμε να αντιληφθούν και εκείνοι οι οποίοι έχουν την επίβλεψη, έχουν την εποπτεία, να αντιληφθούν πόσο σημαντικά είναι τα πράγματα αυτά. Όχι αυτά που πρέπει να κάνουν μόνο οι Βρυξέλλες, αυτά που να κάνετε και εσείς. Να γνωρίζουν και αυτοί λοιπόν τι πρέπει να πράξουν. Αυτή, αυτή την υποστήριξη σας ζητώ. Σας, ευχαριστώ. Επανερχόμαστε στα Εθνικά Κοινοβούλια και δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Τιμό Αρακα από την Φιλανδία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να την προσοχή στο γεγονός ότι η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της διάβρωσης ε, της φορολογικής βάσης αφορά νομοθεσία που δεν είναι από της ε, φορολόγησης δεν είναι κάτι αντίστοιχο με την νομοθεσία για το εταιρικό δίκαιο ή τα λογιστικά. Στην Φιλανδική Βουλή έχουμε σφοδρή ζήτηση για το πώ θα εφαρμόσουμε τη σχετική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κεντρικά ταμιευτήρια αξιογράφων. Επίση, ιδιαίτερα τη ρήτρα που διαπραγματεύτηκε η Φιλανδία και το ζήτησε και το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο άρθρο 38 για να εξασφαλίσουμε το σύστημα που έχουμε στη Φιλανδία, Νορβηγία και άλλες χώρες και που κάνει υποχρεωτική την άμεση ιδιοκτησία των εξωγράφων, ώστε να αναφέρεται στον λογαριασμό του δικαιούχου και να είναι και ε, προσβάσιμη για το κοινό. Δεν θα επισέλθω σε στην πολιτική σύντηση. Πάντως υπάρχει ανησυχία ότι μια τέτοια εφαρμογή νομοθεσία θα αποδυναμώσει την αντίστοιχη νομοθεσία τη Φιλανδία γιατί θα δώσει την ευκαιρία ε, για μεταφορά ε, περιουσιακών σε άλλους ε, λογαριασμούς και σε άλλες χώρες. Κάτι τέτοιο ε, έρχεται σε αντίθεση με τις γενικώ εξέφερνους στόχους Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποκατασταθεί δίκαιη φορολόγηση και σωστά έσοδα στι φορολογικέ αρχέ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, η δημοσίευση του γράφου του Παναμά ενισχύει την έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά υπάρχει κίνδυνο για μείωση διαφάνεια αλλού, σε άλλα σημεία τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ο κανονισμό έχει μια διετή εφαρμογή μέχρι στιγμή, αλλά το όλο περιβάλλον έχει αράξει, έχει αυξηθεί το επίπεδο φιλοδοξία. Γι' αυτό θα πρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ίσως ε, θα πρέπει να κάνουν πιο αυστηρό το θέμα των κεντρικών ταμιευτήριων αξιογράφων ώστε να γίνει περιττή η τωρινή συζήτηση και η εθνική μας εξαίρεση να γίνει ευρωπαϊκός κανόνας γιατί χωρίς διαφανή οικονομικά δεν νοείται αποτελεσματική φορολόγηση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι. Μόνο σου κατάλαβα έχετε δημιουργήσει στη Φιλανδία ένα σύστημα το οποίο εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία ξεωράφων. Και αυτό που μας λέτε είναι, αφού λειτουργεί καλά στις σκανδιναβικές χώρες, γιατί δεν το υιοθετείτε παντού, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανταλλαγή απόψεων που έχουμε υπό αυτή τη μορφή, με αυτές την συναντήσεις μας δίνουν τη δυνατότητα ακριβώς αυτό να κάνουμε. Βεβαίως μπορούμε να συζητούμε τις ευρωπαϊκές προτάσεις, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και επίσης και κυρίως μπορούμε να ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές και ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν όλους, ακόμα και αν το ζήτημα παραμένει εθνική αρμοδιότητα. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Χούμπερτ Φούχς από την Αυστρία. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε και εσείς αξιότιμοι Κυρίες και κύριοι ε, βουλευτέ, είναι βαρύ το φορολογικό βάρος που βαρύνει τους πολίτες και πολύ μεγαλύτερο αναλογικά από αυτό των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Πρέπει επιτέλους να πάψει αυτή η στρέβλωση του φορολογικού ανταγωνισμού. Χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για την βελτίωση της φορολόγησης και της διαφάνειας στην ενιαία αγορά. Αυτά είναι απόλυτα αναγκαία. Και συνεπώς το μέτρο μάλλον συγγνώμη, το πακέτο μέτρων είναι ένα καλοδεχόμενο βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Το βήμα αυτό όμως πρέπει να το ακολουθήσουν και άλλα βήματα, πολλά άλλα βήματα. Για παράδειγμα, μία ενιαία φορολογική βάση που ε, να μην είναι απαραίτητα ε, πανομοιότυπος ο συντελεστής, αλλά να προβλέπει ελάχιστα και ανώτατα όρια. Βεβαίως η φορολογική αρμοδιότητα θα παραμείνει στα χέρια των χωρών μελών. Χρειάζεται, όπως είπα, διαφάνεια, σημαντικό στοιχείο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Διαφάνεια είναι απαραίτητη, πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να είναι δικαιότερη η φορολόγηση. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ε, αποφάσεις tax ruling, τις διαμεθοριακές αποφάσεις tax ruling, δεν επαρκεί ωστόσο. Είναι ένα καλό βήμα, δεν είναι αρκετό. Οι φορολογικές αρχές πρέπει να διαθέτουν πληροφορίες, στη βάση δηλαδή αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και να συνεργάζονται πολύ στενότερα. Πολυεθνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με κύκλο εργασιών και με κέρδη καθώς και με φόρους που πληρώνουν. Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι όμως γνωστά όχι μόνο στις φορολογικές αρχές αλλά και στο ευρύ κοινό. Μόνο αυτό θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στα φορολογικά συστήματα των χωρών. Η προτινόμενη οδηγία για την καταπολέμηση πρακτικών φοροαποφυγής θα πρέπει να διατυπωθεί μεν ουδέτερα, να περιλαμβάνει όμως και την φορολογία πολυεθνικών επιχειρήσεων αποκλείοντας οποιασδήποτε δυνατότητες φοροαποφυγής με την πρόταξη κάποιας θηγατρικής. Επίσης πρέπει να γίνει προσπάθεια να αποξηρανθούν οι φορολογικοί παράδεισοι, αν θέλετε να σας το πω έτσι, απανταχού του κόσμου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ερχόμαστε στις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι από εκπρόσωπο Εθνικού Κοινοβουλίου ε, έχουμε μόνο ένα αίτημα. Ε, ένας μόνο έχει ζητήσει το λόγο. Επομένως, αν κάποιος άλλος θα ήθελε ε, να δευτερολογήσει ή αν κάποιος ο οποίος δεν έχει μιλήσει θα ήθελε να λάβει το λόγο, έχουμε τη δυνατότητα. Μιας και έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας, μπορούμε να ακούσουμε και άλλους σε αυτή τη συνάντηση. Εν τω μεταξύ, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπέρντ Λούκε για την ε, πολιτική ομάδα ICR, τους συντηρητικούς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ζητώ συγγνώμη, είμαι πολύ βραχνιασμένος όπως ακούτε. Δεν ξέρω καν αν θα μπορέσω να ολοκληρώσω αυτά που θέλω να πω. Πού το αρπάξατε το κρυολόγημα στην Κύπρο που είχαμε πάει μαζί. Κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω παρόλα αυτά. Πρώτα, είμαι ιδιαίτερα, ικανοποιη, ιδιαίτερα ικανοποιημένος που φαίνεται... Ε, Λυπούν λοιπόν, πολύ που φαινεται λοιπον πολυ δυστυχως δεν θα μπορέσω να συνεχίσω, λέει ο κύριος Λουκέ. It's a pity. Is there another spokesman for this κρίμα. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος βουλευτής που μπορεί να εκπροσωπήσει αυτήν την πολιτική ομάδα. Δυστυχώς όχι. Μίκαλ Έρε. Εδώ είμαι. Modestement au dernier rang. Donc, euh, Ο κύριος Τόερε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Συγγνώμη, συγχωρείτε, από του φιλελευθέρου. Επιθυμώ να τονίσω ότι τα συμπεράσματα της πρώτης Επιτροπής ΤΑΞ αλλά και του σχεδίου BEPS σημαίνουν δύο πράγματα για μας. Αφενός το θέμα αυτό δεν λύνεται πλέον μόνο από τις χώρες μέλη. Δεν λύνεται πλέον στο εθνικό επίπεδο. Τα είπα αυτά και ο κύριος Πέτερ Σίμων. Η πίστη ότι δήθεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν πράγματα όπως οι επιθετικές tax ruling στο εθνικό επίπεδο αποδείχθηκε ψευδέστηση. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα δεσμευτικό νομικό πλαίσιο από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να αναλύσουν τα εθνικά κοινοβούλια πολύ προσεκτικά εάν αρκούν, εάν αρκεί η εφαρμογή των συστάσεων BEPS για την καταπολέμηση της επιθετικής φορολογικής πολιτικής. Ο συνάδελφός μας από την Βουλή των Λόρδων τόνισε ότι δεν είναι ξεκάθαρη απολύτω η έννοια και η διάκριση μεταξύ των ενιών φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Αυτό μα απασχόλησε πολύ, ομολογουμένω. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα στον ανταγωνισμό είναι εκείνα που πρέπει να εξεταστούν ιδιαίτερω. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, η Ιρλανδία να έχει φορολογικό συντελεστή τη τάξη του 12,5% και να μην τον αμφισβητεί κανεί. Μακάρι να πληρώνονται, να καταβάλλονται φόροι της τάξης του 12,5%. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των ερευνών για τις κρατικές ενισχύσεις βρήκε ενδείξεις ότι ορισμένες επιχειρήσεις κατάφεραν με, νομικό, με ένομο τρόπο τελικά να κατεβάσουν το φορολογικό συντελεστή, τον φόρο που πληρώνουν δηλαδή, σε 0,05%. Εκεί ακριβώς οφείλει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθεί κανείς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θέλουν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνικές να καταλήγουν να έχουν ένα σοβαρό φορολογικό μειονέκτημα. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι το μειονέκτημα αυτό ανέρχεται στο 25-30%. Περισσότεροι φόροι δηλαδή που καταβάλλονται από τις ΜΜΕ. Ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι η ψηφιοποίηση. Στα πλαίσια μιας παγκόσμιας ψηφιακή οικονομίας γίνεται όλο και δυσκολότερο τελικά να εντοπίζει κανείς πού παράγεται η αξία ώστε εκεί να μπορέσει αυτή να φορολογηθεί. Γι' αυτό λοιπόν ζητείτε από την επιστήμη να εξετάσει και άλλους τρόπους, άλλα φορολογικά συστήματα τα οποία θα πρέπει να διαθέτει μια παγκόσμια ψηφιακή οικονομία. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Μάνιξ Βανρέη από τη Γερουσία των Κατοχωρών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ θερμά για την οργάνωση αυτής της συνάντησης. Έτσι μπορούμε να διαβρύνουμε το διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Το πρώτο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνη της στον κόσμο. Ότι δεν πρόκειται να ευοδοθεί το σχέδιο για τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών αν δεν υποστηριχθεί πλήρως και από τα άλλα μέλη του ΩΣΑ και κυρίως τα μεγαλύτερα μέλη του ΩΣΑ, τις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, και την Κίνα, τις μεγαλύτερες χώρες μέλη του ΩΣΑ. Όλοι γνωρίζουμε ότι μία από τις αιτίες των αναντιστοιχειών είναι συνέπεια του φορολογικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το Κογκρέσο δεν έχει καταλήξει σε συνένεση προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς φορολογίας επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ε, οι, οι αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν να αντισταθμίσουν το φόρο γιατί ε, από τη στιγμή μάλιστα που επαναπατρίζουν τα κέρδη τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, οι περισσότεροι βέβαια δεν το κάνουν γιατί υπάρχει δυνατότητα να το αποφύγουν και ένα τρισεκατομμύριο ε, δολάρια βρίσκονται σε δικαιοδοσίες εκτός της εκτός της, των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ολλανδική Βουλή στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, μα είπε ο κ. Ντάιζεμπερκ Θα επιταχύνει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εφαρμόσει τις ε, προτάσεις BEPS. Ε θα την ακολουθήσει όμω ε, η Αμερική, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί αυτό θα είναι παράδοξο. Γιατί αν εμεί έχουμε υψηλότερη φορολογία και αυτό οδηγεί σε λιγότερη, χαμηλότερη φορολογία στις Ηνωμένε Πολιτείε, σίγουρα είναι αντικίνητρο για τις επιχειρήσεις να φορολογούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το πακέτο κατά της φοροαποφυγής, είναι σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Ντέισενμπεργκ για τις συζητήσεις στην Ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων για να τελεσφορήσει το σχέδιο και μάλιστα κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας καλό θα ήταν να περιοριστούμε μόνο στα μέτρα του BEPS, ε της διάβρωσης της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών και να μην επεκταθούμε και σε επιπλέον μέτρα. Ε, τη ρήτρα switchover, ε, τα μέτρα κατά της ε, καταχρηστικής εφαρμογή, παρόλο που υπάρχουν σχετικέ συστάσεις στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, ε, θα θέλαμε να σταθούμε σε τρία επιπλέον σημεία. Πρώτον, διαφάνεια είναι ζωτική σημασία. Συμφωνούμε με τις προσπάθειες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα η Ολλανδική Βουλή δεν είχε εφαρμόσει την, ε, ε τις εκθέσεις αναχώρα από την 1η Ιανουαρίου και έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών με το Μνημόνιο Συνεννόησης ό,τι αφορά τις φορολογίες συμφωνίες τύπου ε, tax ruling και έχουμε αντίστοιχη πρωτοβουλία με 23 αναπτυσσόμενες χώρες για να βελτιωθούν οι ρήτρες τους ε, κατά των καταχρήσεων. Και μία προειδοποίηση καλή η φαλοδοξία, όπως είπε και ο Ισπανός συνάδελφος, αλλά ακόμη καλύτερος είναι ο ρεαλισμός. Γιατί θεσπίζουμε πολλούς νέους κανόνες και κανονισμούς και χρειαζόμαστε τις εφορίες για να τους εφαρμόσουμε στην πράξη. Έχουμε όμως τους απαραίτητους πόρους στις 28 χώρες μέλη για να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα, ιδιαίτερα σε, σε θέματα συνεργασία των φορολογικών διοικήσεων. Γιατί πολύ ωραία η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά χρειαζόμαστε υπαλλήλου ε, εφοριακού που θα εφαρμόσουν τα μέτρα. Ευχαριστώ. Votre dernière remarque est particulièrement judicieuse. Πολύ εύστοχο, ειδικά το τελευταίο σας σχόλιο. Και φυσικά το πρόβλημα ίσως δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και στις 28 χώρες μέλη. Επανέρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την ΚΟΕ το λόγο έχει ο Φάμπιο Ντεμάζη. την Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ αυτά τα Panama Leaks, όπως πιο πριν τα Luxembourg Leaks, μας βοηθούν κατά κάποιο τρόπο. Εγώ ευχαριστώ αυτούς τους καταγγέλλοντες που τα δημοσιοποίησαν αυτά τα πράγματα και που σύντομα θα είναι στα δικαστήρια βέβαια. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν βλέπω μια καθαρτήρια δύναμη ιδίως απέναντι σε γίγαντες όπως Amazon και Google. Ακόμα και αν έγιναν κάποια βήματα μέχρι τώρα, δεν είναι ε, επαρκή. Υπάρχουν ακόμα συμφωνίες αποφυγής της διπλής φορολόγησης και με ευρωπαϊκές χώρες, χώρες μέλη, δηλαδή όπως η Ολλανδία που δεν επιτρέπουν την φορολόγηση σε φορολογικούς παραδείσους. Η πολιτεία Delaware των ΗΠΑ δεν συμμετέχει στην ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχουν και χώρες όπως η δική μου που δεν επιτρέπει την αποκάλυψη στοιχείων των εταιριών γάμματο κυβωτίου όπως λέγονται. Μιλούμε ωστόσο για εγκληματικέ δραστηριότητε. Μιλούμε πίσω από το πλήσιμο του βρώμικου χρήματο κρύβεται ακόμα και η χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Θα συμφωνήσω με τον Βρετανό συνάδελφο που μίλησε πριν. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα σε αυτέ τι εκθέσει των πολυεθνικών ομήλων. Εμένα δεν μου αρέσουν οι μαύρε λίστε. Υπήρχαν μαύρε λίστε και παλαιότερα. Και πρόσφατα ο κ. Μοσκοβισή είπε ότι η Πορτογαλία έχει 75 χώρε σε μαύρη λίστα, η Γερμανία 0. Διερωτώ με πώς θα γίνει, πώς θα συμφωνηθεί τελικά αυτή η μαύρη λίστα. Και σε ό,τι αφορά πάλι τις μαύρες λίστες, ασφαλώς και πρέπει να επιλεγούν λύσεις πολυμερείς, πολύπλευρες. Όμως οι Αμερικανοί για παράδειγμα έκαναν μονομερός σημαντικές ενέργειες απέναντι για παράδειγμα στην Ελβετία, απέναντι στο Λίχτενστάιν. Εγώ νομίζω ότι πέρα από αυτά χρειαζόμαστε και ένα ειδικό ποινικό δίκαιο για επιχειρήσεις που να μας επιτρέψει την έρευνα και την ποινική δίωξη τραπεζών που έχουν διευκολύνει τους πελάτες τους να καταλήξουν σε φορολογικούς παραδείσους. Ασφαλώς και χρειαζόμαστε και ένα ενιαίο φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις στην βάση των πραγματικών τους πεπραγμένων. Δεν μπορούμε να έχουμε επιχειρήσεις όπως η Google με έδρα την Ολλανδία όπου δεν έχει παρά μόνο έναν αυτόματο τηλεφωνητή. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε κοινού συντελεστέ αν δεν συζητήσουμε πρώτα ελάχιστου κοινού συντελεστέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Επενερχόμενοι στου προσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων θα δώσω το λόγο για το Κοινοβούλιο ε, του Βελγίου στην κυρία Βούτερς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων με τα εθνικά κοινοβούλια. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να κλείσουν τα παραθυράκια στον νόμο που επιτρέπουν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις να φοροαποφεύγουν. Κατά την άποψή μου, η ιδανική λύση είναι η υιοθέτηση μέτρων που δημιουργούν μεγαλύτερη διαφάνεια και ενισχύουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Θα πρέπει να ενισχυθεί η διοικητική συνεργασία ε, μεταξύ των κρατών μελών και να εφαρμοστεί το σύστημα των εκθέσεων αναχώρα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ενισχύσει τη διαφάνεια κατά την άποψή μου και γι' αυτόν τον λόγο την υποστηρίζουμε πλήρως. Αυτές οι προκαταρκτικές παρατηρήσεις θα ήθελα να πω και κάποια ε, στοιχεία ακόμα. Δεν πρέπει να ξεχνούμε την κατάσταση στα μικρότερα κράτη-μέλη. Ε, τα μεγάλα κράτη-μέλη συχνά την ξεχνούν, συχνά έχουν διαφορετική άποψη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα μικρά κράτη-μέλη πρέπει να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Και γι' αυτό πρέπει να γίνει και σεβαστή η εθνική αρμοδιότητα ε, της υιοθέτηση της εθνικής φορολογικής πολιτικής ε, με μικρές διαφορές μεταξύ των φορολογικών πολιτικών παραμένει η δυνατότητα ο ανταγωνισμός να είναι χωρίς τρευλώσεις, χωρίς προβλήματα. Επίσης, υποστηρίζουμε πλήρως τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί στο πλαίσιο του ΟΣΑ. Είναι σημαντικό να συνεχιστούν. Αλλά ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αγνοεί τι συμβαίνει και ποιο είναι το πλαίσιο, ε, το παγκόσμιο μέσα στο οποίο ε, λειτουργούμε. σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις ευρωπαϊκές πολιτικές να αποδυναμώνεται η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον στην παγκόσμια οικονομία. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε μια μικρή χώρα όπως το Βέλγιο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Επομένως, όποιο μέτρο και αν υιοθετήσουμε, εξετάζουμε και πρέπει να φροντίσουμε να μην δημιουργεί ε, διοικητικό κόστος, διαχειριστικό άχθο στι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Εάν λοιπόν τα λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ε, συνεργασία, την παραγωγική που είχαμε μέχρι στιγμή για την καταπολέμηση τη φοροαποφύγης. Μην ξεχνάμε και τη σημασία λοιπόν που έχουν τα θέματα αυτά για τι μικρέ χώρε. Συνεχίζουμε λοιπόν με την κύριο Έρνεστ Μαργκάη για τους πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μελετήσαμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την δέσμη μέτρων ε, κατά της ε, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής αλλά πραγματικά έχουμε τεράστιες απώλειες, ε, δισεκατομμύρια ευρώ σε δημόσιους πόρους, σε φορολογικά έσοδα, αλλά φαίνεται αντί να αντιμετωπίσουμε το κύριο πρόβλημα, ε, λαμβάνουμε κάποια βαλωματικά απλώς μέτρα. Ε, ο αρμόδιος Επιτρόπος Μοσκοβισή μίλησε για 70 δισεκατομμύρια το χρόνο, το μισό δηλαδή του κοινοτικού προϋπολογισμού και πολύ λιγότερο από ό,τι αφιερώνουμε στα προγράμματα κοινωνικής συνοχής. Επίσης, ε, φάνηκε η δεδηλωμένη βούληση πολλών ε, χωρών. Μερικά απλώς ε, φορολογούν τα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άλλα δεν ε, φορολογούν τις θηγατρικές εταιρείες, άλλοι προσφέρουν ε, προνομιακές φορολογικές συμφωνίες τύπου tax και άλλοι δίνουν φορολογικούς συντελεστές χαμηλότερες από το μισό και έτσι συγκεντρώνουν ε, τα κέρδη. Μπορούμε να υπολογίσουμε λοιπόν τις απώλειες των των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι τα η απώλεια φορολογικών εσόδων ενώ είναι τρισεκατομμύρια τα κέρδη αυτών των εταιριών που χάνουν ε, ε, που οδηγούν σε απώλεια φορολογικών εσόδων για πολλές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, ενώ οι χώρες με φορολογικούς χαμηλού, χαμηλούς συντελεστές, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, ε, λαμβάνουν πάντα από 50 δισεκατομμύρια. Ε, χώρες χάνουν 120 δισεκατομμύρια και άλλες κερδίζουν. Ε, ε, οι χώρες που έχουν προνομιακά φορολογικά καθεστώτα καρπώνονται 50 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογικά έσοδα. Δεν είναι ακατανόμαστη αυτή η κατάσταση με τέτοιες προτάσεις και με απλέ μαύρε λύσει, πιστεύω ότι θα λύσουμε το πρόβλημα. Μόνο με παγκόσμια λύση και παγκόσμια μέτρα μπορούμε να, θα καταφέρουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Αλλιώ ε, θα συνεχιστεί η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή. Θα έχουμε μεταφορά κερδών ε, στις ε, χώρε με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και όλο και μεγαλύτερη ανισότητα και αδικία. Και ό,τι φεύγει από εμά θα το δούμε στου ίσους Καϊμάν, βερμούδε, στον Παναμά, πάνω από ένα τρισεκατομμύριο είναι η απώλεια φορολογικών εσόδων ε, ετησίως. Γι' αυτό θα πρέπει να κινητοποιηθούμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε στην, ε, στην εύκολη λύση των ε, γράφων του Παναμά. Θα πρέπει να έχουμε πολύ πιο ευρυθή συζήτηση και πολύ πιο ριζικά μέτρα για την συνολική μας εξωτερική στρατηγική πολλές ε, εθνικές βουλές, όπως η Ισπανική, έχουν ζητήσει εξεταστικές υπηρεσίες, εξεταστικές συγγνώμη επιτροπές, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε τελικά με τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο σημαντικό και αυτή είναι η μοναδική προοπτική για τους επόμενους μήνες του κοινοβουλευτικού έργου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επαναρχόμαστε στα Εθνικά Κοινοβούλια και να δώσω το λόγο στο κύριο Ντανιέλ Σέστρασίτς από τη Σουηδική Βουλή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερως για την ε, συμφωνία που υπάρχει μεταξύ μας να πατάξουμε τη φοροαποφυγή, ένα φαινόμενο που μας ε, προβληματίζει και μας ταλαιπωρεί εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια υπάρχει ένα ευρύ ε, φάσμα απόψεων για το πώς θα το επιτύχουμε μπράκτος, αλλά χαίρομαι για την πρόταση αποκατάστασης της διαφάνειας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεμάζη, τον Φάβιο Ντεμάζη, για την ε, πολύ εύστοχη παρουσίαση που μας έκανε. Για την χώρα μου, αλλά και για τις περιφέρειες μας και για τις πόλεις μας, είναι σημαντικό να σταθούμε σε αυτό που είπε ο Σλοβαίνος συνάδελφος. Ότι δηλαδή πολλές χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα απώλειας φορολογικών εσόδων. Και ένα βασικό κενό στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι δεν ε, αντιμετωπίζει πλήρως το θέμα της έλλειψης διαφάνειας. Χρειάζεται και ε, διαφάνεια για το κοινό, για τους δημοσιογράφους, για τους εμπειρογνώμονες, όλοι να έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. Αλλά επίσης σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ποιες χώρες θα υποβληθούν στις εκθέσεις αναχώρα. Το κατόφλι παρά είναι υψηλό. Μιλάμε για 40 εκατομμύρια ευρώ και θα πρέπει να είναι πραγματικά δημόσιες τέτοιες εκθέσεις αναχώρα. Αλλά δεν αρκούν οι ευρωπαϊκές ε, εκθέσεις αναχώρα, ε, δηλαδή μόνο για τις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα αυτές οι εκθέσεις αναχώρα. Και στο μέλλον θα πρέπει να εντείνουμε τις πιέσεις μας προς αρμόδιες αρχές για να έχουμε πραγματικά δημόσια αρχεία και να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι και ποιοι ευνοούνται από τις πολυεθνικές και να διδαχθούμε τέτοια συμπεράσματα από τα έγγραφα του Παναμά. Η κυρία Μπάρμπαρα Κάπελ από το ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καταπολέμηση της φοροαποφυγής καθώς και αυτές οι επιθετικές φορολογικές πολιτικές δεν πλήττουν μόνο την Ένωση αλλά ιδίως και τις χώρες μέλη. Ο στόχος μας πρέπει να είναι κοινός πραγματική αποτελεσματική φορολόγηση των επιχειρήσεων εκεί όπου παράγεται η αξία του προϊόντος τους. Δέχθηκε και πριν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταλήγουν να πληρώνουν 30% και παραπάνω φόρο από ό,τι οι πολυεθνικές. Οι εθνικοί προϋπολογισμοί θίγονται ιδίω από τις επιθετικές αυτές φορολογικές πρακτικές. Μέχρι και 70 δισεκατομμύρια ε, έσοδα από φόρους διαφεύγουν κάθε χρόνο, τα λέει ο αυτά, και καταλήγουν σε φορολογικούς παραδείσους, όπως έδειξε πολύ καθαρά και η υπόθεση του Παναμά. Η πρωτοβουλία του ΩΣΑ με την επικεφαλίδα BEPS είναι σημαντική για την ανακοπή αυτής της παγκόσμιας φοροαποφυγής. Πρόκειται για ένα σχέδιο δράσεως με 15 σημεία και 3 παραμέτρους. Διεθνή συντονισμός για την φορολόγηση των εσόδων των εταιριών, κλείσιμο των φορολογικών παραθύρων και αύξηση της διαφάνειας. 17 από τις χώρες ε, μέλη της Ευρωζώνης έχουν ε, δεσμευτεί να αναλάβουν ε, την εφαρμογή των συστάσεων αυτών. Τώρα και οι Αμερικανοί δέχονται μετά από τα, τη δημοσίευση των εγγράφων του Παναμά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει και σχέδιο για την καταπολέμηση της διεθνούς φοροαποφυγής με τις τρεις αυτές παραμέτρους που ανέφερα προηγουμένως και τις τελευταίες εβδομάδες μάλιστα υπήρξε και ανακοίνωση σχετικά με μητρό διαφάνειας για το country by country reporting για τις ε, πολυεθνικές ε, επιχειρήσεις και για τους φόρους που καταβάλουν αυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και δύο επίκαιρες εκθέσεις που κυκλοφορούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Αφενός το country by country reporting για τις ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις και ομίλους δηλαδή με συνολικό φόρο κύκλου εργασιών άνω των 750 εκατομμυρίων. Αυτό αφορά λοιπόν 6.500 συνολικά επιχειρήσεις. Το ΔΕ ΕΚΟΦΗΝ στις 8 Μαρτίου φέτος συμφώνησε να καταστήσει δεσμευτική την αναχώρα υποβολή εκθέσεων από το 2017 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτά τα μέτρα δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα μια παγκόσμια διαδικτύωση των εθνικών μητρών διαφάνειας και ένα πραγματικό παγκόσμιο δίκτυο που να καταδεικνύει ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από τις εταιρείε γραμματοκιβωτίων. Με την τέταρτη οδηγία για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος προβλέπεται τέτοιο μητρό. Το ίδιο πρέπει να ενοποιηθούν οι μαύρες λίστες, να ληφθεί υπόψη και μια ανάγκη ευθυγράμμισης των προθεσμιών παραγραφής, καθώς και όλες οι σχετικές ρήτρες για ε, φορολόγηση κατά την έξοδο των ε, κερδών και ούτε καθεξής. Τα είπε αυτά και ο Ιταλός συναδελφός μας πριν. Χρειάζεται και μια ε, ξεκάθαρη έννοια, ένας ξεκάθαρος ορισμός της έδρας. Μίλησε ένας συναδελφός μας και για τις ανάγκες της παγκόσμιας ψηφιακής αγοράς. Αυτά επίσης πρέπει να μας απασχολήσουν. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε. Ε, τώρα εκ μέρους της γερουσίας της τσεχικής δημοκρατίας ο κύριος Σέλνεκ. Μου βρίσκεστε αγαπητοί συνάδελφε. Εδώ. λόγω ονόματος της Άνω Βουλής της Τσεχικής Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε ασχοληθεί με ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα φορολόγησης των μεγάλων επιχειρήσεων. Θα συζητήσουμε βέβαια τις ε, προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε βάθος. Γενικά στηρίζουμε πάντως μέτρα κατά της φοροαποφυγής που ασκούν οι ε, μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις, διότι αυτά ζημιώνουν την αγορά, μειώνουν τα κρατικά έσοδα και υπονομεύουν τον ανταγωνισμό. Θέλουμε ωστόσο να τονίσουμε επίσης ότι η άμεση φορολογία είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Παρόλα αυτά και μέσα στα πλαίσια μιας προσπάθειας αντιμετώπισης της φοροαποφυγής, μια συνεργασία στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι όντως επιθυμητή. Θεωρούμε ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιέχουν κατάλληλα μέτρα για, την, ε, τον περιορισμό της φοροαποφυγής και για την διαφυγή εσόδων δηλαδή. Πολλά από τα οποία ήδη εξήγησαν οι προλαλήσαντες συνάδελφοί μου. Θέλουμε να τονίσουμε επίσης ότι δεν προβλέπει η πρόταση χρονικό περιθώριο για την μεταφορά στην εθνική νομοθεσία των σχετικών συστάσεων. Για την τσεχική δημοκρατία τουλάχιστον μπορώ να πω ότι αυτό, η, μετα, η μεταφορά αυτή δηλαδή θα χρειαστεί πολύ χρόνο. Και γι' αυτό θέλουμε να ζητήσουμε περιθώριο τουλάχιστον 24 μηνών. Στηρίζουμε και τη νέα στρατηγική για βελτιωμένη διαχείριση των φορολογικών και στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες και την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βελτίωση της συνεργασίας με διεθνείς εταίρους για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Όπως λέχθηκε ήδη και εμείς συμφωνούμε με την ανάγκη σύνταξης μιας λίστας χωρών που επιτρέπουν τελικά την φοροαποφυγή μέσω επιθετικών φορολογικών πρακτικών σε βάρος άλλων λιγότερο ισχυρών οικονομιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη πρέπει να ασκήσει σημαντική πίεση σε αυτού του φορολογικού παραδείσου και νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο και ένα κατάλογο επιχειρήσεων που εποφελούνται από αυτά τα ευνοϊκά καθεστώτα. Και για τα μπέψε βεβαίω Ευχαριστώ. Η Ευρωβουλευτή κυρία Γκόμε. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες πολύ πιο ενεργά και να ασκούμε πίεση και, στους και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στις κυβερνήσεις μας για να κάνουν αυτό που πρέπει. Και θα αναφέρω ορισμένα παραδείγματα, ορισμένα στοιχεία. Μια κοινή ε, μαύρη λίστα. Μετά, το, στις εκθέσεις αναχώρα. Όχι όμως περιορισμένες όπως αυτές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ε, αναφερόμενες μόνο σε εκείνες τις πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε όλες τις, σε όλες, συγγνώμη, όλες τις πολυεθνικές εταιρείες οπουδήποτε στον κόσμο και αν έχουν την έδρα τους. Ε, γιατί διαφορετικά θα έχει το ακριβώ αντίθετο αποτέλεσμα, θα τι ενθαρρύνει να μεταφέρουν τι δραστηριότητέ του εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, το κατόφλι θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερο από αυτό που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξει πραγματική έλεγχο. Μετά, είναι το κρίσιμο ερώτημα του κατά πόσο θα δημιουργηθεί ένα, μια βάση δεδομένων ε, δημοσίως διαθέσιμη ε, για το, ένα μητρό για τις επιχειρήσεις. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που έχει σχέση μόνο με την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, αλλά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του ξεπλήματος μαύρο χρήματο, ακόμα και της τρομοκρατίας που χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα με τις offshore εταιρείες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το επιτρέπουμε. Έχουμε επιτρέψει τα εγκληματικά συμφέροντα να έχουν υπονομεύσει τις δυτικές μας κυβερνήσεις, δεν έχουμε καταφέρει να προστατεύσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας όπως θα έπρεπε η οδηγία η οποία δεν έχει καν ακόμα τεθεί σε ισχύ, θα πρέπει να ε, επικαιροποιηθεί, γιατί ακόμα και αν δεν έχει εφαρμοστεί, ήδη βλέπουμε ποια είναι τα παραθυράκια της και τα προβλήματά της. Επίσης, κάτι σχετικό. Δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο μητρό αυτό μόνο οι εταιρείε, αλλά επίσης και τα ιδρύματα και τα trust. Όταν είχε συζητηθεί το θέμα αυτό, ορισμένα μέλη του Κοινοβουλίου από το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν δραστηριοποιηθεί έτσι ώστε να μην συμπεριληφθούν τα τραστ. Δεν είναι τυχαίο αυτό, αλλά το ζήτημα είναι κρίσιμη σημασία. Και θα πρέπει να εξαναγκαστεί το Ηνωμένο Βασίλειο να αντιμετωπίσει αυτή την ε, τραγική κατάσταση που έχει επιτρέψει. Αυτό που μετά την δημοσιοποίηση των Panama Papers αναγκάστηκε να κάνει ο πατέρας του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Ιαν Κάμερον, θα πρέπει να εξαναγκαστούν να το κάνουν όλοι οι πολιτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το ζήτημα εδώ είναι πώς αξιοποιούν ε, τέτοιες τράπεζες σε οποιοδήποτε επίπεδο η ευρωπαϊκή πολιτική. Επίσης, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την αγορά ε, των εκτιμάτων και ε, των ακινήτων, γιατί γνωρίζουμε ότι ένα, μια μέθοδος ε, ξεπλήματος μαύρου χρήματος είναι αυτές οι αγορές. Επίσης, στις κάτω χώρες έχουμε μια, ένα φορολογικό παράδεισο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν έχουμε ...16 από 27 εισηγμένες εταιρείες να μεταφέρουν τα κέρδη τους. Ε, Όλα αυτά τα βήματα είναι απαραίτητα εάν θέλουμε να, καταφέρουμε να φτιάξουμε αυτή την ενοποιημένη κοινή βάση εταιρική φορολόγηση. Τέλο. Στη συμφωνία TTIP με τις ΗΠΑ θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ένα κεφάλαιο ε, εκεί που αναφερόμαστε στις άμεσε ε, ε, στις άμεσες επενδύσεις σε ένα, στην υποχρεωτική εφαρμογή του BEPS. Ο πρόεδρος, από ό,τι διαπιστώνω δεν θέλετε να ε, διευκολύνεται τις διαπραγματεύσεις για το TIP. Ο κύριος Αρακά έχει ξαναζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα πάλι το λόγο. Εν μέρη και για να ευχαριστήσω τα αυτιά των διερμηνέων σας να ακούσουν λίγο την ωραία φιλανδική γλώσσα. Βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον εδώ στα ευρωπαϊκά όργανα και γι' αυτό η σημερινή συνάντηση είναι εξαιρετικά σημαντική. Παράδειγμα, η φιλανδική κυβέρνηση δημοσίευσε τους ευρωπαϊκούς στόχους της και εκεί τοποθετείται και για ευρωπαϊκά, υπέρ μάλλον ευρωπαϊκών φορολογικών μέτρων, τα οποία βρίσκει θετική εξέλιξη. Όμως εκφράζει και την ανησυχία ότι τα ευρωπαϊκά φορολογικά μέτρα ενδέχεται να μειώσουν την ανταγωνιστικότητα και των χωρών μελών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα είναι πώς ορίζουμε την ανταγωνιστικότητα. Δεν μπορεί να είναι η πρόφαση αυτό για να αποφευθεί οποιαδήποτε φορολογική προσπάθεια. Οπωσδήποτε προσπάθεια αρρύθμισης των ε, φορολογικών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολίτες δυσανασχετούν με αυτά με αυτούς τους επιθετικούς φορολογικούς σχεδιασμούς των ε, μεγάλων επιχειρήσεων. γιατί θεωρούν ότι παραβιάζουν την ανταγωνιστικότητα των χωρών τους. Χρειάζονται, ωστόσο, μέτρα και, εθνικού, και στο εθνικό επίπεδο. Βεβαίως έχουν και οι επιχειρήσεις τα νόμιμα συμφέροντά τους. Αυτό που κυρίως ζητούν όμως είναι η προβλεψιμότητα των φορολογικών συστημάτων. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποτελέσει ένα κεντρικό στόχο και των αποφάσεων που θα ληφθούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι αν δεν υπάρχει προβλεψιμότητα, δεν θα μπορέσουμε να πείσουμε και τις επιχειρήσεις ότι μακροπρόθεσμα είναι και προς το συμφέρον τους να καταπολεμηθούν οι ε, φορολογικές επιθετικές πρακτικές. Σας ευχαριστώ. Θέλει άλλος κανείς το λόγο παρακαλώ. Γιατί δεν θέλω να στερήσω από κανέναν την ευκαιρία να μιλήσει. Ο Λόρδος Ντέβις, επειδή ασκήθηκαν επικρίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει δικαίωμα να απαντήσει και μετά ο Μιγγέλ Βιέγας. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να δευτερολογήσω. Είμαι ευγνώμων για τα σχόλια των συναδέλφων και τα σχόλιά τους. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κουέστ μία ερώτηση, αν μου επιτρέπει, γιατί βλέπω ότι πολλοί ε, σχολαστικά κρατούσε σημειώσεις όλο το απόγευμα. Στο επεξηγητικό σημείωμα στις οδηγίες για την ε, αποκάλυψη πληροφοριών ε, για φόρο εισοδήματος κάποιων τομέων, στην σελίδα 20, περίπου στη μέση, αναφέρεται ότι στόχος είναι να γίνει ο, έλεγχος, ο δημόσιος έλεγχος για το που καταβάλλεται ο φόρος. Και η πρόταση αυτή αναφέρει δημόσια αποκάλυψη πληροφοριών για το πού καταβάλλεται ο φόρος. Και στην επόμενη σελίδα, στην τέταρτη παραγράφη, αναφέρεται ότι οι πληροφορίες των φορολογικών αρχών δεν είναι προσιτές στο κοινό. Αντίφαση δηλαδή υπάρχει. Τελικά θα είναι δημόσια προσιτές αυτές οι πληροφορίες, είναι ή όχι κύριε Κουέστα. Ελπίζω πάντως ότι στόχος της οδηγίας είναι να καθιστά προσιτές ε, τις πληροφορίες όχι μόνο στις εφορίες αλλά και στο ευρύ Νομίζω ότι είναι απαραίτητο για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο φορολογικό σύστημα γιατί και οι ενδιαφερόμενοι και οι πελάτες ακόμη έχουν δικαίωμα πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε αγαπητοί συνάδελφοι. Όντω ε, τα σημειώνει προσεκτικά όλα αυτά ο κύριο Κουέστ. Κατέγραψε πιστά όλε τι παρατηρήσει και τι ερωτήσει και θα του δώσω σε λίγο το λόγο για να σχολιάσει να απαντήσει. Ο Μίγκελ Βιέγκας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ο τελευταίο μα ομιλητή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποια σύντομα σχόλια. Καταρχήν, ε, είναι πολύ αξιέπαινη πρωτοβουλία οργάνωση αυτής τη συζήτηση, Πολύ χρήσιμη η συζήτηση και κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο ζήτημα που ανακύπτει για το θέμα αυτό είναι να ε, διαπιστώσουμε αν υπάρχει ή όχι πολιτική βούληση για να χτυπήσουμε, να πατάξουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Πολιτική βούληση. Έχουν πολιτική βούληση τα κράτη-μέλη. Γιατί τα, η φορολογία ε, εξακολουθεί να είναι ε, εθνική αρμοδιότητα. Βέβαια, ευτυχώς, υπάρχει αυτή τη στιγμή συνένεση δεν είναι θέμα εναρμόνιση των ε, φορολογικών συντελεστών. Δεν πρόκειται περί αυτού. Το θέμα είναι, γίνεται δεκτή η αρχή με βάση την οποία τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί που παράγονται. Και φυσικά στη συνέχεια με βάση το στυλ, το μοντέλο, την βούληση ε, διακυβέρνησης και τον τρόπο διακυβέρνησης και φορολογικής διακυβέρνησης κάθε χώρας. Υπάρχει όμως συνένεση ως προς την αρχή αυτή, ως προς το στόχο αυτό. Γιατί με όλα αυτά τα σκάνδαλα ε, προσκρούμε στο θέμα. Υπάρχει πολιτική βούληση αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί εργαλεία και μέσα υπάρχουν για να ποινικοποιηθεί ε, η συμπεριφορά αυτή και οι τράπεζες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τους, φορολογικού τους φορολογικούς παραδείσους. Σχεδόν όλες οι χώρες σχεδόν έχουν τους δικούς τους φορολογικούς παραδείσους. Θα πρέπει να διορθώσουμε την ε, ορολογία, γιατί όταν λέμε φορολογικός παράδεισος, έρχεται στο μυαλό μας μια εξωτική χώρα, ενώ στην ουσία οι πιο σημαντικοί φορολογικοί παράδεισοι βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εξαρτάται από τα κράτη-μέλη να διαπιστώσουν αν έχουν, αν διαθέτουν πραγματικά αυτή την πολιτική βούληση να θέσουν ένα τέρμα στους φορολογικούς παραδείσους. Εμείς προτείναμε στην ε, Πορτογαλική κυβέρνηση να σταματήσει, να κλείσει ο φορολογικός παράδεισος της Μαντέρας, αλλά προσκούσαμε σε εμπόδια. Είναι λοιπόν σημαντικό να ευθυγραμμιστούμε όλοι με το στόχο αυτό και να πραγματοποιήσουμε σημαντικά βήματα και να αφήσουμε τις ψευτοδικαιολογίες και τις συστηματικές αναβολές των σημαντικών πολιτικών αποφάσεων που οφείλουμε να λάβουμε. Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η συζήτηση με τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων, γιατί έτσι μπορούμε να διαγνώσουμε αν υπάρχει μια συνένεση ώστε να αποφύγουμε αυτή τη μόνιμη αναβολή στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Ακριβώς επειδή περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει πρωτογείτονα, η γειτονική χώρα. Για μία ακόμη φορά θα πρέπει να εξάρουμε την οργάνωση αυτής της συζήτησης και ελπίζω να πραγματοποιήσουμε και επί της ουσίας αυτά που χρειάζονται πραγματικά να γίνουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Ήταν πραγματικά πολύ ε, πλούσια και μεστή. Θα δώσω το λόγο στο Γενικό Διευθυντή για να δώσει ενδεχομένω κάποιε απαντήσει, να συμπληρώσει κάποιε πληροφορίε, μετά στου δύο συνεισηγητέ για να αντλήσουν τα τελικά συμπεράσματα και θα κάνω και εγώ κάποια σχόλια και παρατηρήσει. Καταρχήν, είναι σαφέ ε, και το επισημάνατε πολύ ότι είχαμε πει και στην εισαγωγή και ο πρόεδρος Ντέιζεμπερ και ο υποφαινόμενος ότι το θέμα αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα. Εσείς θα αποφασίσετε, αγαπητοί συνάδελφοι των Εθνικών Κοινοβουλίων, εσείς θα έχετε τον τελευταίο λόγο. Το, η φορολογία αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Εμείς είμαστε εδώ για να διευκολύνουμε τη συζήτηση μεταξύ σας ώστε να μπορέσετε και εσείς να λάβετε υπόψη την ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση των εθνικών επιλογών που θα πραγματοποιήσετε και επίσης ε, να μεριμνήσουμε ώστε να έχετε όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση και ενημέρωση, κυρίως ε, τις πληροφορίες από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Όλοι συμφωνούμε ότι το ισχύον σύστημα καταλήγει σε κατάφορες αδικίες και πολλοί μας υπενθύμησαν ότι κατά μέσο όρο και είναι Μέσο όρο. Ε, κατά μέσο όρο λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει καταβάλουν ε, υψηλότερου φόρους ε, από τις πολυεθνικές, 30% περισσότερους. Επίσης, η κυρία Βούτερ. ρώτησε αν μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος μιας χώρας ε, είναι ε, σημαντικό κριτήριο και οι μικρές χώρες αν έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από τις μεγάλες. Αυτό μας προβλημάτισε ε, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα κάναμε μια γενική επισκόπηση του συστήματος στο στις ευρωπαϊκές χώρες και πολλές χώρες μας είπαν ότι είναι εύλογο και θεμητό οι μικρότερες χώρες να υιοθετήσουν μεθόδους που δεν χρησιμοποιούν οι μεγάλες χώρες. Αλλά γι' αυτό υπάρχει ακόμη ερωτηματικό, δεν υπάρχει συμφωνία. Και ακόμη και μεγάλες χώρες χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους. Και τώρα, τι εστί μικρή και τι εστί μεγάλη χώρα. Το μέγεθος είναι κριτήριο. Μία χώρα ε, με πληθυσμό πάνω από 10 εκατομμύρια είναι μικρή. Αλλά αν τη συγκρίνουμε το Λουξεμβούργο ή τη Μάλτα, ούτε και αυτό ισχύει. Επαναλαμβάνω λοιπόν, το μέγεθος μια χώρας είναι σημαντικό κριτήριο βαρύνων. Πάντως το βέβαιο είναι ότι ο φορολογικό ανταγωνισμός είναι αναπόφευκτο. Ανάλογα ε, με το πολιτικό κόμμα που αποφέρεται κάθε φορά θεωρείται κάτι τέτοιο θετικό ή αρνητικό. Πάντως ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι αναπόφευκτος και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει όμως να μεριμνήσουμε ότι, ώστε ο φορολογικός αυτός ανταγωνισμός να πληρεί τις αρχές και τους κανόνες ε, που ισχύουν στον ανταγωνισμό και σε άλλους τομείς ώστε σήμερα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω όταν μιλούμε για τη φορολογία και δι, την φορολογία των εταιριών, που είναι το αντικείμενο της σημερινής συζήτηση να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός φορολογικός και όχι αδιαφανής, αθέμητος και άδικος. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε στο κοινό ότι κάποιες χώρες ε, σφετερίζονται φορολογικά έσοδα άλλων χωρών και μάλιστα ε, αυτό το φαινόμενο συμβαίνει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσο δεν το γνωρίζει η κοινή γνώμη επιτρέπεται. Αλλά από τη στιγμή που κοινοποιηθεί αυτό το φαινόμενο και βγει στο φως, είναι αδύνατο να συνεχιστεί. Και μετά το σκάνδαλο του LuxLeaks και μετά τα έγγραφα του Παναμά, θα ακολουθήσουν και άλλα σκάνδαλα φαντάζομαι. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο, διεθνή ο Διεθνής των Δημοσιογράφων που αποκάλυψε τα σκάνδαλα LuxLeaks και Panama Papers ε, και στο οποίο συμμετέχουν χιλιάδες δημοσιογράφοι από πολλές χώρες, ε, συνεχίζει να δραστηριοποιείται και σίγουρα θα ξεσπάσουν και άλλα σκάνδαλα σε άλλες χώρες. Η κοινή γνώμη δεν αντέχει πια άλλες τέτοιες καταστάσεις. Τις ανεχόταν μέχρι τώρα γιατί δεν τις γνώριζε. Οπότε συμφωνούμε ότι η φορολογία είναι εθνική αρμοδιότητα. Συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις φορολογικές αδικίες. Τώρα θα πρέπει να συμφωνήσουμε τι εστί θεμητός ανταγωνισμός, σε συνθήκε ανταγωνισμού και τι εστί διαφανής, θεμητό και έντιμος φορολογικό ανταγωνισμό και δίκαιο επιπλέον. Όλοι συμφωνούμε ως προς τη διαφάνεια και αυτά μα είπε και ο εκπρόσωπο της Φιλανδικής Βουλής, ο κύριος Χάρακα, για το πώς εφαρμόζεται με πολύ αυστηρό τρόπο μάλιστα αυτό στη Φιλανδία. Και αυτό που έδειξε το σκάνδαλο με τα έγγραφα του Παναμά και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο, γιατί το γνωρίζαμε εμένα αλλά τώρα έχουμε περίτρανες αποδείξεις, πολύ πιο κραυγαλές. Αυτό που μας έδειξε λοιπόν το σκάνδαλο των εγγράφων του Παναμά είναι ότι υπάρχει δυνατότητα σε μερικές δικαιοδο... δικαιοδοσίες να δημιουργηθούν ε, πλέγματα εικονικών εταιριών, εταιριών γραμματοκιβωτίων, ε, περίπλοκες ε, νομικές ε, δομές και συστήματα, καταλήγοντας σε λύσεις που είναι νόμιμες σε ορισμένες χώρες και όχι σε άλλες και έχουν πολύ διαφορετικές φορολογικές συνέπειες ανάλογα με τη χώρα στην οποία εμφανίζονται. Και σε μερικές χώρες θεωρούνται διαφανείς και σε άλλες απόλυτα διαφανείς. Είναι λοιπόν ένα τομέα στον οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες ε, και να κάνουμε πιο σημαντικές τομές από ό,τι μέχρι τώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σκοπιμότητα της κατάρτισης μιας μαύρης λίστας των μη συνεργάσιμων, να το πούμε καταφημισμό δικαιοδοσιών. Εδώ υπάρχει διάσταση απόψεων. Όλοι είναι κατά κανόνα υπέρα, αλλά άλλοι έχουν αμφιβολίες και ενδιασμούς γιατί είχαμε μέχρι τώρα μαύρε λίστες, αλλά δεν τι αξιοποίησαμε δεόντω. Ο κύριος Κουέστα μα μας πει πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα πρέπει να συμφωνήσει με τον ΩΣΑ, πώ θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πείσει και τι 28 χώρε μέλη να συμφωνήσουν σε ένα ενιαίο κατάλογο, σε μια ενιαία μαύρη λίστα και να την χρησιμοποιούν με τον ίδιο τρόπο. Γιατί δεν έχει νόημα να έχουμε κοινό κατάλογο, αλλά να οδηγεί σε διαφορετικέ συνέπειε. Ο Μιχαήλ Τόιρερ μας υπενθύμησε ότι μέχρι στιγμής δεν καταλήξαμε σε σαφή απόφαση και λύση για το ποια είναι η διαφορά μεταξύ ε, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Για τη φοροδιαφυγή δεν υπάρχει αφιβολία, είναι αξιόπινη πράξη, είναι παράνομη η ενέργεια. Η φοροδιαφυγή του tax evasion είναι σαφής οι ένομες συνέπειες της φοροδιαφυγής και γνωστές. Τώρα, αν υπάρχει τεχνική διαφορά μεταξύ επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και φοροαποφυγής, tax avoidance, οπότε αν θα πρέπει να καταλήξουμε σε διαφορετική νομική μεταχείριση μεταξύ του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της φοροαποφυγής, tax avoidance, αυτό είναι ένα θέμα στον οποίο για το οποίο δεν καταλήξαμε σε συγκεκριμένη απάντηση, σε συγκεκριμένη λύση. Θα μας πούν τη γνώμη τους και οι συνεισηγητές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διάσταση απόψεων υπήρξε και για το θέμα της εναρμόνισης της φορολογικής βάσης. Αυτό το περίφημο CCCT, το CCTB ή CCTB, δηλαδή κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών ή απλώς ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών. Αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε διαδοχικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει καταρχήν πρόταση επί του ενιαίου ορισμού της φορολογητέας βάσης και αν καταλήξουμε συμφωνία για την ε, κοινή, φορολογική, ε, βάση φορολογίας εταιριών, μετά θα, σε δεύτερο επίπεδο θα δούμε αν θέλουμε να είναι και ενοποιημένοι, γιατί θα έχουμε μεν κοινή βάση φορολογίας εταιριών, αλλά θα έχουμε ίσως διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές. Οπότε ε, διαρωτόμαστε πού θα φορολογείται μία πολυεθνική. Όλοι είπαν ότι η κρατούσα αρχή θα πρέπει να είναι ότι η κάθε εταιρεία θα πρέπει να φορολογείται ανάλογα με το που έχει τις δραστηριότητες και που παράγει κέρδη. Γνωρίζουμε όμως ότι ο ορισμός της οικονομικής δραστηριότητας είναι και αυτός δύσκολος. Με βάση τις συστάσεις του ΩΣΑ ε, συνδυάζουμε τα κέρδη, τον κύκλο εργασιών και τα περιουσιακά στοιχεία. Υπάρχουν όμως πολυεθνικές που οργανώνονται με τέτοιο τρόπο σε κάποιες θηγατρικές τους, που δεν είναι εικονικές αλλά ουσιαστικές, γνήσιες θηγατρικές, με εκατοντάδες ή χιλιάδες εργαζόμενους, ε, διαφορετικά δεν μπορούν να παράγουν κέρδη. Οπότε πού θα καταβάλλεται ο φόρος των κερδών, όχι σε αυτές τις χώρες που δραστηριοποιούνται οι φόρο Και υπάρχει και ένα νέο καινούριο πρόβλημα που δραστηριοποιουνται οι και υπαρχει και ενα πολύ και που θα πρέπει να μας απασχολεί στο θέμα τη της οικονομία, οικονομίας, των ψηφιακών πλατφορμών. Και κυρίως ε, τι γίνεται με τα δεδομένα, γιατί από εκεί προκύπτει ο πραγματικός πλούτος. Δεν φορολογούνται όμως τα δεδομένα αυτά ανάλογα με τα από ποια χώρα προέρχονται. Και επίσης ε, τα έσοδα και τα κέρδη επίσης δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα. Οπότε οι ψηφιακές οικονομίες και οι ψηφιακές πλατφόρμες ε, δημιουργούν ένα νέο λογιστικό πρόβλημα, το πρόβλημα της προστιθέμενης αξίας. Και άρα δημιουργούν και ένα νέο φορολογικό πρόβλημα. Θα πρέπει όμω πρώτα να ακούσουμε του οικονομολόγους. Και από τη στιγμή που οι οικονομολόγοι θα πραγματοποιήσουν την ανάλυση τη προστιθέμενης αξία των ψηφιακών πλατφόρμων, τότε θα δούμε τι συνέπειε θα ε, αντιλήσουν οι εφορίε οι εθνικέ βουλέ. Δηλαδή πρόκειται για έμεση φορολογία. Μερικοί αναφέρθηκαν στο πρόβλημα που δημιουργεί ο ΦΠΑ. Υπάρχουν κάποια στοιχεία λοιπόν και άμεσης ίσως φορολογίας ή θέματα πνευματικη ιδιοκτησία ή άλλα είδη φορολογίας. Ο κύριος Κουέστα σημείωσε ότι ακούσαμε παρατηρήσεις όσον αφορά καθυστερήσεις στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Εδώ και χρόνια έχουμε διμερεί συμφωνίες, αλλά επίσης και την ομάδα εργασία για τον κώδικα συμπεριφορά για την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών. Ήδη από πέρυσι έχει υιοθετηθεί η οδηγία που καθιστά υποχρεωτική την ανταλλαγή πληροφοριών για συμφωνίες τύπου tax rulings. Φαίνεται όμως ότι αυτά τα πληροφοριακά συστήματα, τα συστήματα ανταλλαγής παραμένουν κάπως ε, αργά. Τώρα, όσον αφορά την εφαρμογή εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση των συστάσεων BEPS, ε το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτέ ή αν θα πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, όπω για παράδειγμα στην ε, πρόταση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το switchover, το οποίο έχει δημιουργήσει κάποιε ε, αντιγνωμίες. Και όπως είπε και ο ε, εκπρόσωπο του Ουρανικού Κοινοβουλίου στην αρχή και πολλοί συνάδελφοι το είπαν, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να συνεργαζόμαστε με άλλους διακυβερνητικούς οργανισμούς. Και όπως σας είπα, ε, στα μέσα Μαΐου στο Παρίσι, στην έδρα του ΟΣΑ, διοργανώνουμε μια κοινή συνάντηση, στην οποία θα παρευρεθεί μια ε, αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας. Επίσης, αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας θα παρευρεθεί ε, θα, θα, θα ε, μεταβεί στις ΗΠΑ για να συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών και με τον Κογκρέσο. Είχαμε ανταλλάξει και παλαιότερα όμως απόψεις μαζί τους και πολύ ευγενικά μας είχαν απαντήσει ότι αυτά τα πράγματα δεν μας αφορούν, it's none of our business. Από τότε όμως τα πράγματα άλλαξαν μια μεταστροφή. η οποία προκλήθηκε από το γεγονό ότι η φαρμακοβιομηχανία Pfizer αποφάσισε να ε, μεταφέρει την έδρα της στην Ιρλανδία. Κάτι το οποίο δημιούργησε αντιδράσεις στις ΗΠΑ σε ένα ζήτημα το οποίο το συζητάτε στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας στην Αμερική. Η, η κυβέρνηση έλαβε μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να περιορίσουν τέτοιου τύπου πρακτικές και πιθανότατα να μην επιτρέψουν στη Pfizer τελικά να μεταφέρει την έδρα της. Αλλά ταυτόχρονα το Κογκρέσο και τα δύο σώματα και τον ε, των αντιπροσώπων και η Γερουσία έχουν αποφασίσει να ξεκινήσουν ακροάσεις και στο πλαίσιο αυτών των ακροάσεων να δώσουν μεγαλύτερη ε, έμφαση, να εξετάσουν πιο ενδελεχώς τις προτάσεις του ΩΣΑ. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και με αυτή την ευκαιρία θα συναντηθούμε με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας για να τους παρουσιάσουμε αναλυτικά τις ευρωπαϊκές θέσεις. Δηλαδή το γεγονό ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια εφαρμογή των ε, συστάσεων BEPS σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την ε, πρωτοβουλία και επίσης στο ε, εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν είμαστε αφελείς με οποιαδήποτε τέτοια εφαρμογή συστάσεων δεν θα πρέπει να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα κανενός εκ των δύο. Σας ευχαριστώ κύριε Κουέστ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους παρεμβάντες για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Θα ομαδοποιήσω τις απαντήσεις μου γύρω από τρία θέματα. Πρώτα την ανάγκη ανάληψης δράσης, το επίπεδο ανάληψης δράσης και τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Για την ανάγκη ανάληψης δράσεως πολλοί νομίζω και από διάφορες ε, γωνιές φώτισαν την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της απώλειας εσόδων. Συζητήσαμε ποια είναι η πραγματική ε, φορολόγηση, ποια είναι η φορολογική βάση και ούτω καθεξής. Ενδιαφέρουσα συζήτηση και αν τα συνδέσω αυτά με τις διάφορες προτάσεις που έχουμε υποβάλει για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και το πρώτο σύνολο προτάσεων που έχουμε σε αυτή τη δέσμη μέτρων για την φοροαποφυγή είναι σχεδιασμένο για να αντιμετωπίσει κάποια από τα προβλήματα αυτά. Και ίσω να έρθω στο δύσκολο πρόβλημα των ορισμών. Δεν ξέρω αν νομοτεχνικά θα σα ικανοποιήσω απόλυτα. Από τη μια μεριά έχετε την, φορο αποφυ... την φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή που είναι ποινικό κολάσιμο, αδίκημο, σε αυτά, αδίκημα συμφωνήσαμε σε αυτά όλα. Από την άλλη μεριά έχουμε την φόρο αποφυγή. Αυτή είναι και, η έννοια αυτή είναι και στην καρδιά τη συζήτηση που έχουμε τώρα. Κάποιες μορφές φοροαποφυγής μπορεί να είναι και νόμιμες, υποθέτω. Η πιο ουδέτερη από αυτές είναι η εκμετάλλευση κάποιων κινήτρων για επενδύσεις κτλ. Εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εφόσον αυτές είναι διαφανείς και είναι διαθέσιμες σε όλους. Μετά όμως μπαίνετε λίγο σε μια θεά ζώνη και εκεί παίζει ένα ρόλο η εκμετάλλευση κάποιων ε, παράθυρων της φορολογικής νομοθεσίας που ενδέχεται να είναι καταχρηστική. Και η επιθετική φορολογική πρακτική είναι όταν οδηγείται στα άκρα αυτή την προσπάθεια φοροαποφυγής, εκμεταλλευόμενος, η εκμεταλλευόμενη η ε, επιχείρηση δηλαδή, πράγματα όπως ε, εξαιρέσεις από, από διπλή φορολόγηση, από ε, επιστροφές φόρων που έχουν διπλά φορολογηθεί και Αυτά είναι και ζητήματα δικαιοσύνης στην βάση του ανταγωνισμού. Αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε εδώ είναι η φορολόγηση να είναι έντιμη, δίκαια, ισόρροπη και σε ίσο πεδίο ανταγωνισμού. Να αποφύγουμε λοιπόν τα παράθυρα και τα κενά στην νομοθεσία που επιτρέπουν σε ορισμένους να αποφεύγουν να πληρώνουν τη δίκαιη φορολογία. Κάτι άλλο που έπαιξε ρόλο στη συζήτηση ήταν η σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών και η διαφάνεια. Είναι χρήσιμο να ακούει κανείς την στήριξη των διαφόρων προτάσεων που βρίσκονται στη διαδικασία της ε, έγκρισης, σχετικά δηλαδή με την ανταλλαγή πληροφοριών. Έχουμε ήδη σύστημα, το οποίο εγκρίθηκε πέρσι, ανταλλαγής πληροφοριών για τα tax ruling. Έχουμε συστήματα που προβλέπουμε τώρα για την υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Αυτό όμως είναι μονάχα μεταξύ φορολογικών αρχών. Έχουμε και πρόταση πρόσφατα για μια υποβολή αναφορών εκθέσεων αναχώρα που θα είναι δημοσιοποιημένες πλέον, θα είναι δημόσιο κτήμα δηλαδή. Αυτή την ε, πρόταση θα την εξετάσουμε. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι κοινό κτήμα. Συζητούνται πολύ εδώ από ό,τι είδα και η κάλυψη το κατόφλι αυτής της πρότασης. Τώρα οι προτάσεις πλέον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν μπει στον πολιτικό χώρο και θα πρέπει να γίνουν βέβαια συζητήσεις έτσι ώστε να βρεθεί μια δίκαιη ισορροπία που να επενδύσει την πρόταση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε ότι υπάρχει στήριξη από παντού υπέρ της διαφάνειας αυτής και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει τον ρόλο της για την εφαρμογή αυτών των διεθνών συμφωνιών. Πολλή συζήτηση έγινε και για μαύρες λίστες. Είτε θέσατε το ερώτημα, λειτουργούν, αποδίδουν, δεν αποδίδουν. Είναι ευαίσθητο, είναι ακαθόδες το θέμα. Και θα δούμε ότι, μάλλον κάναμε μια πρόταση ήδη από τον Ιανουάριο, για να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διασφαλίσουμε μια προώθηση μιας σωστής φορολογικής διαχείρισης παγκόσμια με τη συνεργασία και με την καταχώρηση σε καταλόγους εταιριών που δεν συνεργάζονται. Και τώρα πάμε να αποκαταστήσουμε ένα σύνδεσμο ανάμεσα στην πρόταση εκείνη του Ιανουαρίου και στην ε, υποβολή εκθέσεων αναχώρα, που θα γίνει δημόσια όπως υποτίθεται, όπως έλεγε η πρόταση προ δύο εβδομάδων. Να συνδυαστούν τα δύο αυτά πράγματα δηλαδή και να έχουμε ένα σύστημα εγγραφής σε καταλόγους όταν θα αρχίσει να ισχύει και η υποχρέωση της αναχώρας υποβολής εκθέσεων. Ο διακόπτη πρόεδρος, με συγχωρείτε. Τι κυρώσεις θα προβλέπονται, υποθέτω ότι θα προτείνεται μια κοινή κύρωση για τις δικαιοδοσίες εκείνες που θα μπουν σε μαύρες λίστες. Θα έχουν βέβαια μια κακή φήμη πρωτίστως, αλλά αυτό αρκεί. Ποιες θα είναι ας πούμε οι νομικές και πρακτικές συνέπειες της εγγραφής κάποιου στο μαύρο κατάλογο. Κύριος Κουέστ. Για να απαντήσω σύντομα μπορώ να πω ότι μάλλον η διαδικασία που προτείνουμε είναι να συζητηθούν στην ομάδα του κώδικα διοντολογίας πρώτα ποιες χώρες θα πρέπει να εγγραφούν στην λίστα και να συμφωνήσουν οι χώρες μέλη που εκπροσωπούνται στην ομάδα αυτή ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Η πρώτη λοιπόν απάντηση θα πρέπει να είναι ότι η πρώτη κύρωση είναι ας πούμε η δημόσια ανακοίνωση και έτσι λοιπόν η έκφραση δυσαρέσκειας απέναντι στη συγκεκριμένη χώρα. Και αυτό είναι αρκετά αποτελεσματικό γιατί έχουμε δει χώρε οι οποίε έχουν μπει στι λίστε να είναι εξαιρετικά διατεθειμένε να πράξουν τα πάντα για να βγουν. Δεν έχουν μπει όλε τι λίστε. Ορισμένε ναι, ορισμένε όχι. Είναι μία πτυχή λοιπόν του προβλήματο αυτή. Και θα πρέπει μετά να ξεκαθαρίσουμε ποιε θα είναι οι επιπτώσει στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο εθνικό επίπεδο. Λαμβάνοντα υπόψη βέβαια και την αρχή τη επικουρικότητα. Αυτό είναι ωστόσο ο στόχος της πρότασης. Το πώς θα το χειριστούμε αυτό. Ναι, αλλά φανταστείτε ότι μια τράπεζα που έχει μια θηγατρική σε μια δικαιοδοσία που υπά... περιλαμβάνεται στη μαύρη λίστα ή έχει ε, οικονομικές συναλλαγές με μια τέτοια δικαιοδοσία θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε ότι δεν θα δικαιούται μια τέτοια τράπεζα να δραστηριοποιείται πλέον στην Ευρώπη. Θα ήταν απλούστατη η συνέπεια. Μπορεί να είναι κάπως ομές αυτές οι αποφάσεις, αλλά το Κογκρέσο όχι μόνο λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις, αλλά τις εφαρμόζει και στις δικές τράπεζες όταν έχουν εμπορικές συναλλαγές με άλλες χώρες. Για διαφορετικούς λόγους. Αν δεν ε, υιοθετήσουμε τόσο αυστηρές ε, κυρώσεις, τότε θα μείνουν όλα στη θεωρία. Δεν θα παραμείνουν στη θεωρία. Ο στόχος, ο πρωταρχικός στόχος είναι να εξασφαλίσουμε χρηστή φορολογική διακυβέρνηση και να επιλύσουμε το πρόβλημα στην πηγή, ώστε να μην χρειαζόμαστε τέτοια μαύρη λίστα με δικαιοδοσίες. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε ε, έναν αποτελεσματικό κατάλογο ώστε να ε, ξέρουν, να ξέρει η γνώμη ποιες, για ποιες δικαιοδοσίες πρόκειται και να ξέρουν και αυτές τι πρέπει να κάνουν για να αποφύγουν το πρόβλημα. Και φυσικά θα περιλάβουμε κυρώσεις, αλλά είναι θέμα επικουρικότητας, επαφείται στα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι τμήμα της πρόκλησης, γιατί εργαζόμαστε ταυτόχρονα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Και τέλος, το θέμα του ανταγωνισμού. Ή της ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει κατά την υποβολή αυτών των προτάσεων να προασπίσουμε και να διαφυλάξουμε την ανταγωνιστικότητα των εταιριών μας. Οπότε, μήπως θα πρέπει απλώς να εφαρμόσουμε το BEPS ή να εφαρμόσουμε πρώτα το, την αμυγή πρόταση BEPS και να έχουμε ξεχωριστά κάποιες άλλες πτυχές πέραν του BEPS. Η προσέγγιση μας είναι σφαιρική, εφαρμόζει τη, με ολοκληρωμένο τρόπο τη, το σχέδιο δράση BEPS, αλλά λαμβάνει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της εσωτερικής αγοράς και νομίζω ότι είναι πιο σωστό να το συμπεριλάβουμε σε μια νέα πρόταση που την υποβάλαμε τον Ιανουάριο και με αυτή την βάση θα θέλαμε πρόοδο. Παραμένει το θέμα όμως αν θα γίνει δεκτή αυτή η πρόταση, να μείνουν σε μια νέα οδηγία τα δύο θέματα ή θα τα διαχωρίσουμε σε δύο ξεχωριστές προτάσεις όπως πρότειναν κάποιοι ε, βουλευτές. Αλλά αυτό είναι πολιτική απόφαση. Και συνεχίζεται η συζήτηση για το θέμα αυτό υπό την αιγύδα της Ολλανδικής Προεδρίας και ίσως έχουμε ήδη το Μάιο. Πάντως όπως και να έχει, ελπίζουμε όλες οι πτυχές, οι μεμονωμένες πτυχές πρόταση να εγκριθούν, γιατί είναι όλες σημαντικές για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα θέματα. Αν παρέλειψα κάτι θα μου το επισημάνετε, με βέβαιος. Ο, Γε, ο Γέπε. Το τελικό λόγο τον έχουν οι δύο συνεισηγητές μας. Γέπε Κόφοντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την πολύ επικοδομητική συζήτηση που είχαμε. Πιστεύω ότι από τη συζήτηση καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη συζήτηση. Για να ε, διευκρινίσουμε ε, περισσότερο τις έννοιες. Για παράδειγμα, τι ακριβώς σημαίνει φοροαποφυγή και τι ακριβώς σημαίνει ε, επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός τι επίσης σημαίνει ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, τι ακριβώς σημαίνει υγιής ανταγωνισμός. Όλες αυτές τις λέξεις, όλες αυτές τις έννοιες πρέπει να τις συζητήσουμε περισσότερο, να τις ορίσουμε καλύτερα. Πρέπει τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουμε ότι θα, υπάρξουν, θα υπάρξουν ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού και είναι κανόνες για όλους και επίσης να φροντίσουμε να μην κλέβει η μία χώρα τα φορολογικά έσοδα της άλλης. Το λέω με τρόπο ξεκάθαρο, αλλά η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η διάβρωση της φορολογικής βάσης της Ευρωπαϊκής συνολικά, αλλά επίσης και ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών. Αυτό είναι προκλητικό για τους ε, πολίτε μα. Αυτό είναι πρόκληση επίση, να το βλέπουν να σημαίνει, αυτό είναι πρόκληση επίση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, όταν αναγκάζονται να πληρώνουν περισσότερου φόρου από τι ε, μεγάλε πολυεθνικέ. Είναι κάτι το οποίο υπονομεύει την επιχειρηματικότητα. Δεν επιτρέπει σε νέε εταιρείε να, να δραστηριοποιηθούν. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το του οίκου μα. Επίση, όσον αφορά τι φορολογικέ συμφωνίε τύπου tax rulings, ανταλλάσσουμε πληροφορίε για αυτέ αλλά δεν θα έπρεπε να είχαμε ε, περισσότερες ε, πληροφορίες και για άλλα ε, συστήματα, άλλα μορφές εταιρικής χρήσης εταιρικών μορφών που ίσως να χρησιμοποιούνται για φοροπροφυγή. Πιστεύω ότι έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε σε αυτό το τομέα. Επίσης, ας μην ξεχνούμε ότι βρισκόμαστε μέρος ενός μιας παγκόσμιας οικονομίας, όπου το κεφάλαιο κυκλοφορεί ελεύθερα. Επομένως, δεν μπορούμε να αγνοούμε την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γνωρίζουμε ότι 3 εκατομμύρια δολαρίων έχουν ξεφύγει από τις Ηνωμένε Πολιτείες και αυτό το έχουν επιτρέψει το Αμερικανικό Κογκρέσο. Μπορεί να μην είναι κάτι παράνομο, αλλά αυτό δεν αρκεί. Αντιστοιχεί σε αυτό που ακούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα. Διαπιστώνω ότι υπάρχουν κενά και παράθυρα στην ε, νομοθεσία και αυτά πρέπει να κλείσουν. Αυτό δεν έχει γίνει λοιπόν ακόμα. Και πολλά άλλα. Για παράδειγμα για την πραγματική κυριότητα. Εδώ δεν είναι μόνο ζήτημα ε, διαφάνειας, αλλά επίσης να μην είναι το σύστημα το, της δόμησης μιας εταιρεία υπερβολικά περίπλοκο. Ακριβώς το αντίθετο με αυτό που είδαμε στις εταιρείε που αναφέρονται στα έγγραφα του Παναμά. Ε, τι νόημα θα είχε να γνωρίσουμε ποιο είναι ο κύριο ο, ο ιδιοκτήτη μια εταιρεία, εάν τελικά πίσω από αυτόν τον ιδιοκτήτη κρύβεται ένα άλλο και ένα άλλο και το όνομα δεν μα λέει τίποτα. Πρέπει λοιπόν αυτού του τους κανόνες να τους εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο. Το ζήτημα των εκθέσιμων αναχώρα το έχουμε συζητήσει πολλέ φορές. Κατά την άποψή μου, το πιο απλό, το πιο ξεκάθαρο θα ήταν να ε, εφαρμόσουμε τους ε, ίδιους κανόνες με εκθέσεις αναχώρα που να καλύπτουν όλες τις πολυεθνικές εταιρείε, όχι μόνο τις τράπεζες. Έχουμε κανόνε για τι τράπεζε να, εφαρμόσουμε, να εφαρμόσουμε τους ίδιους κανόνες για όλες τις πολυεθνικές. Και αυτό βέβαια πρέπει να συζητηθεί πιο διεξοδικά. Ακούγοντας τη συζήτηση σήμερα, διαπιστώνω ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη στην πρωτοβουλία της Επιτροπής για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής αφενός και την πρωτοβουλία BEPS του ΩΣΑ αφετέρου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και επίσης να μας επιτρέψει να έχουμε ηγετική θέση στην παγκόσμια συζήτηση που γίνεται ε, και στους G20 και στον ΟΣΑ. Για παράδειγμα, όταν ξέρουμε ότι ο κ. Κάμερον έχει κάνει μια συμφωνία και ε, δικιά του δικαιοδοσία ίσως να μπορείτε να χρησιμοποιείτε για σχεδιασμό ή φοροαποφυγή. Πιστεύω. Ε, μάλλον έχει κάνει συμφωνία η οποία του επιτρέπει να έχει πληροφόρηση σε σχέση με ε, τέτοιους, τέτοιες δικαιοδοσίες. Τη ίδια πληροφόρηση θα πρέπει να έχουν και τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη. Αντιστοίχω, αν οποιοδήποτε κράτο μέλο καταφέρει να συλλέξει πληροφορίε για έναν φορολογικό παράδεισο, για μια τέτοια δικαιοδοσία, θα πρέπει να την ε, μοιράζεται με όλε τι υπόλοιπε. Είναι κάτι το οποίο το διαπιστώσαμε με τι διάφορε διαρροέ του τελευταίου ε, χρόνου ε, ότι οι εταιρείε εκμεταλλεύονταν ακριβώ αυτή τη ροή πληροφοριών που δεν υπήρχε. Μόλι έχουμε ξεκινήσει όπω έλεγα υπάρχει η απαιτούμενη ε, πολιτική δυναμική, αλλά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε η δημοσιοποίηση των εγγράφων του Παναμά και πέρασε οι πρώτες δύο εβδομάδες και σταμάτησε η αγανάκτηση, εντάξει, πέρασε αυτό. Και φαίνεται σαν να τελματώνει η συζήτηση. Τελικά που καταλήγουμε πιστεύω ότι έχουμε εμεί κοινή, από κοινού ευθύνη να συνεχιστεί η δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά. Όπω σήμερα κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Γιατί οι πολίτε μα έχουν αντιληφθεί ότι η πρώτη αντίδραση, η πρώτη συζήτηση μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων του Παναμά εντάξει, ολοκληρώθηκε και ζητούν το επόμενο βήμα και θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ένωση συνολικά και τα κρατημέλη πολύ πιο γοργά από ό,τι συνήθω τα καταφέρνουν. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Γιέπε. Μικάλη. Σας ευχαριστώ και εγώ ε, και σας κύριε Πρόεδρε και σας αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Μένει να ε, προσθέσω τρία πράγματα. Πρώτον, είχα την εντύπωση ότι οι συνάδελφοι των Εθνικών Κοινοβουλίων εκτίμησαν την ε, δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και ως ένας εκ των δύο συνεισηγητών θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους εθνικούς βουλευτές που έκαναν τον κόπο να έρθουν εδώ στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν μαζί μας τα θέματα αυτά. Δεύτερο θέμα είναι ότι ακούστηκαν πολλά σχόλια προς στήριξη των προτάσεων και ιδεών που έχουμε γράψει εμείς εδώ στην ημερήσια διάταξή μας από την Γαλλία, από την Πολωνία τάχθηκαν υπέρ του συστήματος CCCTB, της κοινή ενοποιημένη δηλαδή Φορολογικής βάσεως επιχειρήσεων, που είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που προωθεί το Κοινοβούλιο. Ε, πολλοί ζήτησαν περισσότερη διαφάνεια. Ε, όντως ε, και αυτό είναι από τα πιο σημαντικά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην νομοθεσία που προχωρεί προς εφαρμογή, υπάρχουν και κάποιες διαφορές ανάμεσα στο αν θα πρέπει οι αρμοδιότητες να τοποθετηθούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο ή αν θα πρέπει να διατηρηθούν στο εθνικό. Εγώ θα ήθελα να προτείνω να μην προκαλέσουμε αντίθεση στα θέματα αυτά. Ως ένας από τους δύο συνεισηγητές θεωρώ ότι ένα από τα πιο σημαντικά που διαπιστώσαμε είναι ότι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που πλήττει, ζημιώνει τις χώρες μέλη. Άρα η επίλυση του προβλήματος είναι προς το συμφέρον των χωρών μελών. Όμως είναι προφανές ότι δεν μπορούν να το χειριστούν μόνες τους οι χώρες μέλη. Χρειάζεται κάποιο είδους διεθνή συνεργασία. Είναι θετικό λοιπόν το ότι ο ΩΣΑ η G20 επιλαμβάνονται του θέματος. Όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να παίξει ένα κρίσιμο ρόλο στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος. Ιδίως έχοντας υπόψη ότι έχουμε και μια ενία αγορά που προβλέπει και την ελευθερία κινήσεως κεφαλαίων. Και από την άποψη αυτή λοιπόν υπάρχει ένα στέρεο επιχείρημα που ζητεί από τις χώρες να βρουν μια κοινή προσέγγιση με, το, με, το, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να βρουν δηλαδή κοινού τόπου για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή. Μάλιστα, σα ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Λαμασούρ. Νομίζω ότι πράγματι εργαστήκαμε καλά. Στην βάση αυτή τη πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα συνεχίσουμε τον προβληματισμό μα καθώς και τις εργασίες μας δίνω ραντεβού σε όλες και όλους σας όσοι μπορείτε να προσέλθετε στο Παρίσι στις 2 Μαΐου για την άλλη αυτή κοινοβουλευτική διάσκεψη που είναι και πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσέλθουν πολλές δεκάδες κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι από όλες τις υπήρους του κόσμου. Σε ό,τι αφορά τις εργασίες, τη εργασίες της δικής μας ειδική Επιτροπής ΤΑΞ θα απολύξουν σε προτάσεις που θα γίνουν τον Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενδιαμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδεχομένω θα εγκρίνει η ίδρυση νέας εξεταστικής επιτροπής για τα προβλήματα που προέκυψαν από τη δημοσίευση των εγγράφων Παναμά και όπως είπε ο κ. Ντάιζενμπεργκ, η Ολλανδική Προεδρία έχει θέσει σε αυτήν στόχο να καταλήξει σε πολιτική συμφωνία επί του συνόλου της δέσμης για τον αγώνα κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης μέχρι τον Ιούνιο πληροφοριακά για τους εθνικούς βουλευτές σημειώνω ότι εργαζόμαστε στα πλαίσια και άλλης κοινοβουλευτικής επιτροπής, της Επιτροπής Οικονομικών, πάνω σε μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας σχετικά με τις απάτες που στρέφονται γύρω από τον φόρο προσθέμενης αξίας. Μέγα πρόβλημα για όλους τους εθνικούς μας προϋπολογισμούς. Βρισκόμαστε στην φάση, βρισκόμαστε μάλλον ενώπιον μιας πραγματικά ε, διεξαγωγής απάτης στην, ε, σε βάρος του ΦΠΑ, θα έλεγα βιομηχανικής κλίμακας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να εναρμονιστούν κάποια πράγματα Ήδη για τις ε, χώρες που ήταν από τις ιδρύτριες της Ένωσης η φορολογική βάση του ΦΠΑ είναι εναρμονισμένη εδώ και 40 χρόνια. Όμως δεν έχουμε μπορέσει να βάλουμε τέλος στις απάτες αυτές και είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν. Σας ευχαριστώ και πάλι όλες και όλους για την συμμετοχή σας. Σας εύχομαι καλή επάνωδο στις πατρίδες σας και ελπίζω να σας ξαναδώ σύντομα για συζητήσεις και για το θέμα αυτό αλλά και για άλλα. Έρετε συνεδρίαση, θα επανέλθουμε στην ίδια αίθουσα. Οι συντονιστές, καθώς και οι συγητές και σκιώδεις συγητές, για να ακούσουμε τους εκπροσώπους των νησιών Καϊμάν. Έρετε συνεδρίαση.